Γεια σας, καλώς ορίσατε στην Επιτροπή την Οικονομική και Νομισματική. Πρώτα απ' όλα θα εγκρίνουμε τα πρακτικά, την, έγκρι, την ημερήσια διάταξη μάλλον. Πάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής μας της ενεδριάσεως 26 Φεβρουαρίου αν δεν έχετε πρόβλημα, τα πρακτικά θεωρούνται εγκεκριμένα. Πάμε στο επόμενο σημείο της ανακοινώσεις του Προέδρου. Στο CR3 έχουμε διορθωτικό. Μετά έχουμε το θέμα της βαθμολόγησης των, ε, της 16 Φεβρουαρίου Έχουμε λοιπόν διορθωτικό για τον κανονισμό και την οδηγία που το ετοίμασε η Διεύθυνση Νομοθετικών Πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 261 του εσωτερικού κανονισμού. Λοιπόν, έχουν ε, στις 8 Απριλίου δοθεί τα κείμενα στα αγγλικά και σε όλες τις γλωσσικές εκδοχές στις 10 Απριλίου. Εν τη απουσία αντιρρήσεων, τα διορθωτικά αυτά κείμενα θα υποβληθούν στο Κοινοβούλιο θα ανακοινωθούν στην Ολομέλεια και θα θερθούν ως συγκεκριμένα εκτός αν υπάρξει πολιτική ομάδα που υποβάλει κάποιο σχετικό αίτημα και ο αναγκαίος αριθμός μελών να ζητήσει να τεθεί ψηφοφορία. Διορθωτική του ΤΟΥΠΑ συμφωνία με το Συμβουλίο όσον αφορά τον κανονισμό της εποπτείας της οικονομικής προσωπικής έκθεση του κ. Γκοζές και την έκθεση της κ. Φερέιρα η Ολομέλεια θέτησε τη θέση της το Φεβρουάριο του Φεβρουαρίου, μάλλον στη δεύτερη, στις 2 Μαρτίου, 12 Μαρτίου 2013. Σύμφωνα με το άρθρο 294, 4 για τον κανονισμό λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωσης αν το Συμβούλιο εγκρίνει θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, η νομοθετική πράξη θα υιοθετηθεί στη διατύπωση που αντιστοιχεί στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μετά από έγκριση στην Ολομέλεια, το κείμενο τώρα έχει βρει την τελική του μορφή μετά την συνεργασία με τους νομο, ε, νομοσομαθείς νομικούς, με τους εισηγητές κλπ. Ανακοινώνω ότι βάσει αυτών των πράξεων διορθωτικό σύμφωνα με το άθρο 2.16 εσωτερικού κανονισμού του Κοινοβουλίου έχει ετοιμαστεί για τα δύο κείμενα και έχει διανεμηθεί στα μέλη. Το σχέδιο αυτό διορθωτικού κειμένου θα ανακοινωθεί στην ενακτήρια στην έναρξη της Ολομελίας του Απριλίου. Μετά την ενημέρωση όσον αφορά το τριμερή διάλογο, μετά το δεύτερο πολιτικό διάλογο, τριμερή διάλογο για τα φορολογικά, επετέθη συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο ε, το μήνα Μάρτιο. Είναι, είμαστε κοντά σε τελική συμφωνία. Εκτός από τις οριζόντιες ε, ρυθμίσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο συμφώνησαν στις 10 Απριλίου σκιώδης. Σχόλια μπορούν να υποβληθούν μέχρι 20 Απριλίου. Αν συμφωνείτε, πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι η δια... εκ νέου διαβούλευση ε, που λαμβάνει η χώρα με την Επιτροπή Αναδιαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 70 στις 20 Μαρτίου του 2013 καταλήξαμε στις κελεφουλικές απαιτήσεις ειδικό κανονισμό και οδηγία σε συμφωνία επί Ιρλανδικής Προεδρίας με τη συμμετοχή του Επιτρόπου Μπαρνιέ. Παραμένουν κάποιε εκκρεμότητε μετά από τι διαπραγματεύσει με την Δανέζικη, Κυπριακή και Ιρλανδική Προεδρία. Η πολιτική συμφωνία επετεύθη 20 μήνε αφού έκανε πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2011. Η Κορεπέρα επιβεβαίωσε αυτή τη συμφωνία, την επικύρωσε στις 27 Μαρτίου. Η επιστολή έχει διανεμηθεί ε, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής μαζί με το σχέδιο ενοποιημένου κειμένου. Θα ήθελα να έχουμε αναδιαβούλευση με την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 70. Και θα δώσω το λόγο στον εισηγητή για να σχολιάσει. Ο κύριος Καράς λοιπόν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε άλλο. Θα σας παρακαλούσα να σημειώσουμε την ε, επιστολή και να ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα μετά από τη συζήτηση στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κάρα. Θα ήθελα τώρα να σας ζητήσω για να προσθεθεί χειρός, να επιβεβαιώσουμε την πρόταση της Επιτροπής να καταθέσουμε το κείμενο στην ε, Ολομέλεια. Υπέρ, κατά, αποχές, το συμπεφωνημένο κείμενο, λοιπόν, θα κατατεθεί προ ψήφιση στην Ολομέλεια του Απριλίου. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε λίγα λεπτά γιατί αναμένεται να ξεκινήσουν 9.30 οι ψηφοφορίες. Να περιμένουμε λοιπόν λίγα λεπτά ώστε να προσέλθουν ε, και άλλοι συνάδελφοι για να μπορέσουμε να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Ευχαριστώ. Καλημέρα και πάλι περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Τις ψηφοφορίες συγκεκριμένα. Πρώτα απ' όλα έκθεση Σάντσες Πρεσέδο για την αιτήσια πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτα απ' όλα να ελέγξουμε τις κάρτες, να βάλετε πρώτα απ' όλα βέβαια τις κάρτες και να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. Ένας ακόμη. Πέρας ψηφοφορίας. Ωραία, είμαστε εντάξει, ευχαριστώ. Περνάμε λοιπόν αυτής αμέσω στις ψηφοφορίες και ξεκινάμε... Α, τι γίνεται. Λοιπόν, να ξανακάνουμε μια δοκιμαστική. Ένα δοκιμαστική, ε. Lo paramos, no? Πέρας της δοκιμαστικής. Τώρα λειτουργεί καλά το σύστημα. Ωραία, λοιπόν, περνάμε τώρα στις ψηφοφορίες και ξεκινίζουμε με την έκθεση Πρασέδο. Συμβαστική ε πρώτα απ' όλα δεν καλύπτει την τροπολογία 33. Θα ψηφιστεί χωριστά η 33. Έχουμε λοιπόν στην 3α τμηματική ψηφοφορία πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Νομίζω πρέπει να ελέγξουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα. Παράγραφος 4. The ε, Εντάξει, κύριε Σφάμπα. Θα επαναλάβουμε και πρέπει να προσθέσουμε και την ψήφα του μέλους του ECR που δεν έχει ηλεκτρονική κάρτα. Αν δεν σας πειράζει λοιπόν επαναλάβουμε το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 3α Η ΕΣΥΑΡ ψηφίζει κατά από ό,τι βλέπω. Τρεις ακόμα παρακαλώ. Ψηφίστε. Δύο. Ωραία. Πέρας λοιπόν τώρα της ψηφοφορίας. Με την ECR έχουμε 14 ε, υπέρ 15 κατά, άρα απορρίπτεται. Παράγραφος 4 τώρα, πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ψήφι περ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Στην παράγραφο 4α πρώτο τμήμα, ψήφι περ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ψήφι υπέρ. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 33. Ψήφι υπέρ. Υπέρ. Δεν βλέπω κανέναν. Ψηφίζουμε την τροπολογία 33 παρακαλώ. Έχει ζητηθεί χωρίς η ψηφοφορία. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 34. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 35. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 43. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική F που δεν καλύπτει την τροπολογία 52, η οποία και θα ψηφιστεί χωριστά. Λοιπόν, περνάμε στι ψηφοφορίε κατά τμήματα. Παράγραφο 9 καταρχάς, ψήφι υπέρ, κατά, απόχέ. εγκρίνεται. Στην παράγραφο 10, πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ψήφι υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, ψήφι υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική F. Α, όχι, κάνω λάθος. Τι κάνουμε, ψηφίζουμε ή δεν ψηφίζουμε εδώ. Όχι. Λοιπόν, όχι, ψηφίζουμε. Συγγνώμη, αλλά υπήρξε ένα πρόβλημα. Λοιπόν, ψήφι υπέρ της F. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 50 ψηφιπέ Κατά αποχές απορρίπτεται. 52 ψηφιπέ Κατά αποχές απορρίπτεται. Όχι, ελέγχουμε. Ελέγχουμε την τροπολογία 52 ηλεκτρονικά. ECR is voting. Οι CR ψηφίζουν κατά. Λοιπόν, εγκρίνεται 16 ψήφοι υπέρ, 14 κατά. Παρακαλώ, εσείς ψηφίσατε υπέρ, είπατε. Δεν αλλάζω το αποτέλεσμα. Ωραία, 17 ψήφοι υπέρ, 14 κατά. Τροπολογία 54, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε την 54. Μάλιστα. Η ΣΥΑ ψηφίζει υπέρ και ο Σκούτα κατά. Άρα τι γίνεται. Δύο ακόμη παρακαλώ να ψηφίσετε. Πέρας ψηφοφορίας. 16 υπέρ, 16 κατά. Άρα απορρίπτεται. Συμβαστική G. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα τη παραγράφου 12. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική G. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολή 69. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική H. Κατά τμήματα. Παράγραφος 14, πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 14 β. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 σι γάμα, πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 15α. Ψήφι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τώρα συμβαστική H, που στροποποιήθηκε υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική I κατά τμήματα. Παράγραφος 20. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική I όπως τροποποιήθηκε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. IA συμβιβαστική. Ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 89 ψήφι υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε. Τροπολογία 89 άρχεται η ψηφοφορία. Ένας ακόμη δεν έχει ψηφίσει. Πέρας. 19 υπέρ, 11 κατά. Εγκρίνεται η τροπολογία 89. Και πηγαίνουμε στην συμβαστική IB. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 92. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 93. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε την τροπολογία 93. Κύριος Γκέπελης, κατά. Μάλιστα. Λοιπόν, 14 ψήφοι υπέρ, 19 κατά απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 94 ψήφοι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική I, C, ψήφι υπέρ. Τι θέλετε, θέλετε να ελέγξουμε την 94. Ωραία. Ελέγχουμε. Πέρας ψηφοφορίας. 17 υπέρ 13 κατά. Επομένω εγκρίνεται η τροπολογία 94. Συμβιβαστική IC. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 104, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 105, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, θα ελέγξουμε την τροπολογία 105. Άρχεται η ψηφοφορία. 18 υπέρ, 15 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 106. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβεβαστική J. Χωριστή. Μάλλον κατά τμήματα. Παράγραφος 24. 2. Τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική J. Όπως τοποποιήθηκε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τραν 22. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τραν 31. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική K. Περ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική L. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Employment 2, ψήφι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Employment 10 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Ή να ελέγξουμε καλύτερα. Να ελέγξουμε. Employment 10. Ένας ακόμη δεν έχει ψηφίσει, παρακαλώ, να ψηφίσει. Πέρας ψηφοφορίας. 16 υπέρ, 16 κατά. Άρα απορρίπτεται. Employment 17. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική M. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική A. Α. Περ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική B. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική C υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική D υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το κείμενο όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά. Είναι ένας που δεν έχει ψηφίσει. Α, εγώ ήμουνα. Πέρας 32 ψήφοι υπέρ, μία κατά και μία αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν το κείμενο και συγχαίρουμε τον εισηγητή κύριο Σάντσεφ Πρέσεφ. Συγχαρητήρια Αντολίνη. Και περνάμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία. Σχέδιο ψηφίσματος από την Προεδρό μας, Άρουν Θα ψηφίσουμε παράγραφο 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 2α. Νέα. Ψήφι υπέρ. 2α. Περ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Ψήφι υπέρ. Κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 3α. Συγγνώμη, τροπολογία 2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Όχι. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε την τροπολογία 2. Λοιπόν, το αποτέλεσμα. 16 ψήφοι υπέρ, 15 ψήφοι κατά και 2 αποχές. Επομένως, απορρίπτεται. Και τι κάνουμε τώρα, ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 4. Ψήφι υπέρ. Εγκρίνεται. Παράγραφος 5 υπέρ κατά, αποχές πρόεδρος λέει πρώτα, κατά αποχές. Εγκρίνεται, παράγραφος, τροπολογία 3, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. Την τροπολογία 3, αρχίζει ψηφοφορία. We close the vote. Πέρας ψηφοφορίας. 16 υπέρ, 18 κατά. Ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε το αρχικό κείμενο. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. 21 ψήφι υπέρ και 13 ψήφι κατά. Επομένως εγκρίνεται. Τροπολογία 4 ψήφι υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 6β, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος, μάλλον τροπολογία 8, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε την 8, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 18 υπέρ 14 κατά. Εγκρίνεται επομένως. Παράγραφος, μάλλον τροπολογία 5. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 7. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε σε τολικές σκέψεις τα recitals. Α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σ. Γ. Δηλαδή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δ. Δ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στα citations, στις αιτιολογικές αναφορές. Το ένα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το δύο, παρακαλώ τι είπατε. Να τα ψηφίσουμε unblock, μαζί όλα λοιπόν τα citations, στις αιτιολογικές αναφορές. Ωραία, συμφωνούμε. Υπέρ, παρακαλώ ποιοι είναι, κατά, αποχές εγκρίνονται. Τώρα ψηφίζουμε το κείμενο όπως τροποποιήθηκε, ηλεκτρονικά. Αρχιέται η ψηφοφορία. να προσθέσουμε και δύο ψήφους υπέρ και αποτέλεσμα 23 ψήφοι υπέρ, καμία κατά και 11 αποχές. Συγχαίρουμε λοιπόν την πρόεδρό μας. Και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ολοκληρώσει εδώ τις ψηφοφορίες και μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα, στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι το σημείο 7. θέσπιση ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα του φόρου των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Εξέταση του σχέδιο έκθεση τη κυρία Άννη Ποδηματά. Να δώσω αμέσω το λόγο στην κυρία Ποδηματά. Thank you ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα θα συζητήσουμε το σχέδιο έκθεσης του Κοινοβουλίου για την για την αναθεωρημένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιβολή ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών για 11 κράτη-μέλη, σύμφωνα με την διαδικασία συνεργασίας Μιλάμε για... Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συμμετέχοντες για την επικοδομητική συνεργασία ως τώρα, κοιτώντας ε, τους βουλευτές που συμμετέχουν στη συζήτηση αυτή, κοιτώντα την αίθουσα, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να ξεκινήσει από την αρχή η συζήτηση από το πρώτο σημείο, γιατί θεωρώ ότι τα βασικά στοιχεία σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών έχουν ήδη συζητηθεί και το Κοινοβούλιο έχει εκφράσει τις απόψεις του, τις τοποθετήσεις του σε διάφορες περιστάσεις. Άρα, Εισαγωγικά θεωρώ ότι είναι σημαντικό να σας υπενθυμίσω ότι τα 11 κρατημέλη που κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή απέφθηναν μια επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζήτησαν η αναφερμένη πρόταση να είναι το δυνατόν ε, εγκύτερη στην αρχική πρόταση, δηλαδή με ευρύ πεδίο εφαρμογής αφενός και κατά δεύτερον σημείωσαν την ανάγκη να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποφευθεί η μετεγκατάσταση. Θεωρώ ότι και οι συγητές και οι πιο πολλοί εξημών συμφωνούν με τους στόχους που έχουν τεθεί και λοιπόν στην έκθεσή μας αυτούς τους σκοπούς θα επιδιώξουμε να πετύχουμε. Ιδιαιτέρως θα ήθελα να καλωσορίσω ένα βασικό στοιχείο στην αφαιρημένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το γεγονός ότι στην πρόταση αυτή ένα από τα βασικά στη σημεία που συμπεριλαμβάνεται είναι η εισαγωγή της αρχής έκδοσης issuance principle ως, τελευταίο, ως τελευταία λύση δηλαδή επιβολή φόρων επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και μέσων που έχει εκδοθεί σε ένα μέλος της επικράτειας του συμμετέχοντος κράτους μέλους. Αυτό είναι σημαντικό θεωρώ για να είναι πολύ στεναρό το μέτρο του φόρου και να μην υπάρχει κίνητρο για την μετεγκατάσταση. Επίσης να θυμόμαστε ότι η πρόταση αυτή είναι η πρώτη απόπειρα να επιβληθεί ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και αυτό συνδέεται με τη συζήτηση για την στενήτερη συνεργασία, τη βαθύτερη συνεργασία σε τέτοια ζητήματα. Ξέρουμε ότι αυτό έχει μια συγκεκριμένη ορμή σε ό,τι αφορά το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ως γενική λοιπόν προσέγγιση στη δεύτερη αυτή έκθεση. Θεωρώ ότι σκοπός μας θα πρέπει να είναι η ενίσχυση του πλαισίου του FTT. Να προσπαθήσουμε να κλείσουμε κάποια κενά. Να εφαρμόσουμε κάποια μηχανισμούς για να αποφύγουμε την αντικατάσταση τη φυγή, την φοροδιαφυγή. Να είναι αποτελεσματική η εφαρμογή και ομοιόμορφη στα 11 κράτη-μέλη, τα οποία σε πρώτη φάση θα κινηθούν προς την κατεύθυνση επιβολής του φόρου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις βασικές μας προτάσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συμπεριέλαβε στην αναθεωρημένη πρόταση της την αρχή του, της ιδιοκτησίας, ownership principle, το οποίο συμπεριλαμβανόταν στην προηγούμενη έκθεσή μας. Μία αρχή η οποία, από ό,τι ξέρετε, ε, προέρχεται από την επιτυχία του stamp duty στο Ηνωμένο Βασίλειο, του φόρου τελών. το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατείνεται ότι δεν μπορεί να συνδεχθεί στην οδηγία η αρχή της ιδιοκτησίας, γιατί δεν ε, έχουν όλα τα κράτη-μέλη τις διοικητικές ικανότητες να τον εφαρμόσουν. Ωστόσο, τα κράτη-μέλη τα οποία πραγματικά θέλουν να εφαρμόσουν τον φόρο επί των χρηματοδοτικών συναλλαγών, θεωρώ ότι φέρουν ευθύνη να δημιουργήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει. Η αρχή της συντεκτησίας δεν θα πρέπει να θεωρείται ως βάρος, αλλά ως ένα σημείο κλειδί, προκειμένου να μην φτάσει σε τέτοια ύψη φορο αποφυγή, ώστε να είναι μη εφικτή. Ε, τώρα, ένα θέμα για την αρχή της έκδοσης. Στην αρχή βέβαια σας είπα ότι η προσθήκη της αρχής ε, έκδοσης από την Επιτροπή είναι κάτι που καλωσορίζουμε. Η εξαίρεση των παραγόγων θεωρούμε ότι ανοίγει ένα παραθυράκι το οποίο ενδεχομένως να βλάψει το σύνολο του μηχανισμού του φόρου γιατί είναι κατά της αρχής ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλες οι αγορές, όλοι οι φορείς και όλα τα μέσα. Και νομίζω ότι, πολύ φοβάμαι ότι δημιουργεί κίνητρα προκειμένου οι συναλλαγές να κινηθούν από τις διαφανείς αγορές προς την κατεύθυνση των OTC, των αγορών OTC. Θα πρέπει να έχει ευρύ πεδίο εφαρμογής, ακόμα και με τη συμπερίληψη ε, των παραγωγών OTC, προκειμένου να είναι ίση η όρια ανταγωνισμού για όλους τους φορείς σε όλες τις αγορές, σε ό,τι αφορά την αρχή του της διαμονής. Θεωρώ ότι θα, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής τα υποκαταστήματα νέων ε, ιδρυμάτων σε τρίτες χώρες, προκειμένου να καλύπτονται και αυτά από τους φόρους. Τώρα, να στραφώ στο πώς θα διασφαλίσουμε την μέγιστη εναρμόνιση και αποτελεσματικότητα των ε, μηχανισμών ίσπραξης. Νομίζω ότι το έχω τονίσει και στο παρελθόν. Πρόκειται για ένα κλειδί, ένα σημείο κλειδί για την επιτυχία του μηχανισμού του φόρου. Τα συμμετέχοντα λοιπόν κράτη-μέλη. θα ήθελα να τονίσω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν στο έπακρο όλη την αιμοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την συλλογή και την πράξη φόρων σε μη συμμετέχοντα κρατημέλη και θα ήθελα να τονίσω ότι τα κρατημέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν υποχρέωση διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας με την οδηγία 2011-16 και για αμοιβαία βοήθεια για θέματα που έχουν να κάνουν με τέλη φόρους και άλλα μέσα με την οδηγία 24 2010 σε ό,τι αφορά τις τρίτες δικαιοδοσίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες για να διευκολυνθεί η εισπράξη του φόρου. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώσει τον ορισμό των μη συνεργαζόμενων περιφερειών και ανάλογα να προσαρμόσει και τα μέτρα για την φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή. Επίσης, προτείναμε να δημιουργηθεί μια ε, επιτροπή ευθυτή που θα αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών, από την ΕΣΜΑ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία θα συζητά τακτικά πώς μπορεί με τον βάλτιστο τρόπο να ε, αξιοποιήσει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την ε, φορολογία και θέματα συνεργασίας ε, όπως ορίζονται από διεθνείς οργανισμούς από το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο ΑΣΑ κτλ. Στο ίδιο πνεύμα σκοπεύουμε να προτείνουμε πράξεις κατά εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις σε θέματα ίσπραξης να είναι δεσμευτικές, υποχρεωτικές αυτές οι πράξεις κατά εξουσιοδότηση και οι εκτελεστικές πράξεις. Αυτά λοιπόν, συνάδελφοι, είναι τα βασικά στοιχεία της ε, έκθεσης, του σχεδίου έκθεσης. Προσβλέπω στα σχόλιά σας, στις παρατηρήσεις σας και προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας, ιδιαίτερως με τους κοιόντες εισηγητέ. για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η, η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 23η Απριλίου. Αυτά από δικιά μου από πλευρά. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστούμε κυρία Ποδηματά. Σα ευχαριστούμε που μα ε, βοηθάτε και που αναφέρετε και το χρονοδιάγραμμα. Και τώρα να διώσω το λόγο στου Κιώδη. Ο κ. Μαρκάρα από το ΕΛΚ καταρχά. Πρόεδρε, συνάδελφοι, καταρχά να ευχαριστήσω την εισηγήτρια Είμαστε ένα, μια καλή συντονισμένη ομάδα σε πολλά ζητήματα. Και νομίζω ότι η έκθεση που μας έχει κατατεθεί και η οποία μας ε, παρουσιάστηκε και προφορικά και την έχουμε μπροστά μας και γραπτά αποτελεί μια πολύ καλή βάση για τις περαιτέρω αντιπραγματεύσεις και για μια ευρεία συνένεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τέσσερα σημεία θα ήθελα να αναφέρω. Πρώτον, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η ενισχυμένη συνεργασία 11 κρατών μελών είναι η τέταρτη καλύτερη λύση. Στόχος θα πρέπει να είναι να συνεργαστούν όλοι τα κράτη-μέλη και να υπάρξει ένας καθολικός φόρος. Θα πρέπει να πούμε ότι εμείς ως στόχος, ως στόχο θεωρούμε την επιβολή ένας τέτοιου φόρου. Η έκθεση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση τη διατύπωση θεωρώ ότι θα πρέπει να τη δυναμώσουμε όμως λίγο και θα σας υποβάλω σχετικές προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Δεύτερη παρατηρήση. Ο φόρος επί των συναλλαγών για πολύ κόσμο αποτελεί ένα θέμα πολιτικής ε, τάξεως και όχι ένα θέμα μόνο ε, που σκοπό έχει να συλλέξει χρήματα. και μου λείπει λίγο αυτό το θέμα της πολιτικής τάξεως. Γι' αυτό θεωρώ ότι οι εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές θα πρέπει να φορολογούνται πιο πολύ από τις χρηματιστηριακές συναλλαγές. Τα κράτη-μέλη μπορεί να είναι πιο αυστηρά, αναφέρει η έκθεση. Θεωρώ ότι και στον ίδιο την νομοθεσία θα πρέπει να ορίζουμε ότι οι εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές θα πρέπει να φορολογούνται πιο, ε, με πιο ψηλό συντελεστή από τις υπόλοιπε. Αυτό δεν είναι θέμα διακριτικής ευχέρειας. Δεν μπορεί το κράτος μέλος να κάνει θέλει, γιατί πρέπει να το κάνει. Τρίτη παρατηρήση. Τα έσοδα από το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα πρέπει να εισραίουν στον ε, προπολογισμό της Ένωσης εάν θέλουμε να υπάρχει αυτή η προστιθέμενη αξία. Εγώ είμαι σαφώς κατά της εισρωής στους εθνικούς προϋπολογισμούς, για να μειωθεί δηλαδή η εθνική συνεισφορά στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. De facto δηλαδή δεν θα υπάρχει ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι επειδή είναι μόνο 11 τα κρατημέλη, αλλά η αρχή θα πρέπει να είναι σαφής. Εφόσον είναι ήδη, ήδη πόροι, θα πρέπει να προστίθενται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και όχι να αντικαθιστούν εθνικές συνεισφορές. όπου έτσι κι αλλιώς υπάρχει ένα θέμα σε ό,τι αφορά τη συνεισφορά που ορίζεται στο 1,42% από την συνθήκη. Τέταρτη παρατηρήση. Θα πρέπει να είναι ευρύ το πεδίο εφαρμογή, αλλά κάποιε λεπτομέρειε θα πρέπει να κάτσουμε να τις σκεφτούμε. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά ε, τι συναλλαγέ Intergroup. Το CED4 ε, σε ό,τι αφορά την ρευστότητα των τραπεζών συμφωνήσαμε και ψηφίσαμε ότι είναι βασικό θέμα της Βασιλείας 2 και του CED4 αυτό της ε, ρευστότητας των τραπεζών. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια συνοχή και μια, μια μορφία με την νομοθεσία αυτή. Και γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε να συζητήσουμε το εξής. Να εξαιρεθούν οι συναλλαγές εντός της ομάδας, όπως ε, συμβαίνει ήδη σε κάποιες χώρες, όπως στη Γαλλία, στην Ιταλία. Θα ήθελα επίσης να είναι ενιαία η επιβολή του φόρου. Ακούω από πολλά κράτη-μέλη ότι χαίρονται που επιβάλλεται αυτός ο φόρος, γιατί έχουν ε, ε, περιθώριο λιγμού προς τα πάνω τα κρατημέλη. Αυτό όμως θα προκαλέσει στρεβλώσεις του τεγωνισμό. Εγώ θέλω να μην ε, είναι έτσι τα πράγματα γιατί θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη στρέβλωση από ότι υπάρχει ήδη σήμερα. Και προς την κατεύθυνση λοιπόν αυτή θα υποβάλω πέντε τροπολογίες. Ευχαριστώ και πάλι την Ανυποδήματα για την έκθεσή της. Okay. Sean, Otmar, I will give... Ευχαριστώ. Στον κύριο Τερμό θα δίνω το λόγο για την άλλη Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια για τη δουλειά που έκανε. Ε, βρισκόμαστε στη συζήτηση αυτή για τον φόρο χρηματοστηρικών συναλλαγών μετά πολλές συζητήσεις και δεν είναι εύκολο για την ομάδα μου το θέμα διότι η ομάδα μου ε, δεν, έχει, δεν κινείται όλοι στο ίδιο μήκος ε, κύματος, υπάρχουν αποκλίνες απόψεις. Υποστηρίζω προσωπικά την ιδέα ότι πρέπει να σεβαστούμε την απόφαση κάποιων κρατών μελών που αποφάσισαν να υπάρξει αυτός ο φόρος. Είναι πολύ φιλελεύθερη θέση. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη, 11, που θέλουν αυτή τη λύση και το σέβομαι. Όμως, θα ήμουν υπέρ του φόρου αυτού εάν εξετάζαμε προσεκτικά τις λεπτομέρειες. Κάτι που θα αναφέρω αργότερα, θα σχολιάσω αργότερα. Καταρχάς, είμαι υπέρ υπέρ του ότι τα εισοδήματα από το φόρο αυτό των, των συναλλαγών να πηγαίνουν στους ίδιους πόρους του προϋπολογισμού. Το κοινοβούλιο δεν θα ήταν κανονικό κοινοβούλιο αν δεν είχε εξουσία συλλογής των φόρων, ίσπραξης των φόρων. Θα προχωρήσουμε βελτιώνοντας τον έλεγχο που μας ζητούν να κάνουμε ε, οι πολίτε, Αν έχουμε σαν κοινοβούλιο τους ιδίου πόρου και πρέπει να λογοδοτούμε για τους πόρους. Εγώ είμαι υπέρ του να πάνε τα χρήματα αυτά μέσα στο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκής Ενώσης και αν κατάλαβα σωστά αυτά που είπε ο κύριος Ότμαρ Κάραξ είμαι υπέρ του, αυτά, του ότι αυτά τα χρήματα, τα νέα χρήματα που θα αυξάνουν τον προπολογισμό της Ένωσης από το φόρο αυτόν να μην εξαλείψουν αυτόματα τις μεταφορές που κάνουν τα κράτη-μέλη αυτές τις μέρες. Προσωπικά, προσωπική άποψη, να έχουμε αύξηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ενώσεως παρά να μείνει στο ίδιο επίπεδο ο προϋπολογισμός. Σχετικά με αυτό, και είναι η προσωπική μου άποψη, δεν είναι η θέση της ομάδας των φιλελευθέρων, ε, αυτή είναι η άποψή μου που εξέφρασα. Έχω κάποιες κόκκινες γραμμές, κάποια όρια, διότι ο φιλελευθερισμός Όταν οι φιλελεύθεροι βλέπουν περισσότερους φόρους και παρεμβάσεις, φιλοσοφικά φοβόμαστε. Φοβόμαστε απροσδόκητες συνέπειες και στρεβλώσεις που μπορεί να επιφέρει ένας ε, νέος φόρος. Η προσωπική μου κόκκινη γραμμή και όριο και νομίζω ότι μου στηρίζει και η ομάδα μου είναι η εξή. Να αποφύγουμε αρνητικές συνέπειες όσον αφορά τα συνταξιωτικά ταμεία ε, και στις αγορές για το δημόσιο χρέος. Οι χρηματοστικές αγορές είναι πολύ διαφορετικές είμαι υπέρ ασύμετρης προσέγγισης. Προσωπικά δεν θέλω να δω τις αγορές του δημοσίου χρέους να, μειωθού, να, να δουν να μειωθεί η ρευστότητά τους μετά την φορολόγηση αυτή και επίσης και για τα συνταξιωτικά ταμεία έχω παρόμοια θέση. Πρέπει να κάνουμε διάκριση όσον αφορά αυτούς τους τομείς. Συμφωνώ με την εισηγήτρια στην τροπολογία 6, όπου η εισηγήτρια λέει ότι ζητάμε περισσότερο δυναμισμό όσον αφορά το φόρο χρηματοστικών συναλλαγών, FTT. Ο χρηματοστικός τομέας έχει μεγάλες δυνατότητες καινοτομίας. Υπερασπίζομαι αυτή τη θέση, πάλι προσωπικά μιλώντας, συμφωνώ με αυτή την τροπολογία, αλλά έχω ανησυχίες όταν αφορά την τροπολογία 7 που λέει ότι ίσως πολλά κράτη-μέλη μπορούν να ζητήσουν υψηλότερο ποσοστό, να εφαρμόσουν υψηλότερο ποσοστό. Αυτό για μένα δεν είναι καλή ιδέα. Είμαι πιο κοντά στη θέση του συγητή του Ελκ Ότμαρ Κάρας που λέει ότι καλύτερο θα ήταν να μην έχουν διαφορετικά ποσοστά φορολόγησης στα διάφορα κράτη-μέλη. Εγώ θα ήμουνα προσωπικά πάντα υπέρ εναρμονισμένου φόρου, διότι θυμηθείτε ότι ο φόρος εισοδήματος ξεκίνησε σαν 1%. Και είπαν μην ανησυχείτε, θα φορολογήσουμε τα εισοδήματα. Μην ανησυχείτε, θα είναι μόνο 1% και βλέπουμε ότι έχουν φτάσει 40, 50, 60% τα ποσοστά του φόρου εισοδήματος σε κάποια κράτη-μέλη. Άρα σαν φιλελεύθερος ανησυχώ όταν από την αρχή καλούμε τα κράτη-μέλη να το κάνουν αυτό, ότι μπορούν να αυξήσουν το φόρο. Έχω ανησυχίες λοιπόν όσον αφορά την τροπολογία 7. Και τέλος υπάρχουν κάποιες τεχνικές φύσεως λεπτομέρειες όπως τροπολογία 16. Μιλάμε για μεταφορά διάφορων τίτλων. Ε, πρέπει να το μελετήσω το θέμα προσεκτικά για διευκρίνηση. Ευχαριστώ, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολύ για τη δουλειά που κάνατε και θα υποβάλουμε τροπολογίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Ραμόν. Εκ των Πρασίνων, ο κ. Μπέσετ, ο σκιώδης εισηγητής, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε ανήκω σε πολιτική οικογένεια η οποία εδώ και 20, 25 χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, πολεμά ε, για την εισαγωγή αυτού του είδους φόρου στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό τοπίο. Με πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση υποδεχόμαστε λοιπόν και υποστηρίζουμε αυτό το πρώτο βήμα που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. πέρα από διακηρύξεις και λόγια. Ε, και είναι μια κίνηση αξιόπιστη. Για μας είναι προφανές ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει μια απάντηση εξαιρετικά θετική στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στις τροπολογίες της κυρίας εισηγήτριας. Μια θετική απάντηση, θα έλεγα μάλλον ενθουσιώδη απάντηση σε αυτό το φόρο, ε, διότι η πολιτική σημασία του στο κλίμα αυτό της κρίσης ε, και της ύφεση ε, στην Ευρωπαϊκή Ήπερο είναι πάρα πολύ, κάτι πολύ σημαντικό. Είναι ένα διαφορετικό μήνυμα που αποστέλλεται σε μια κοινή γνώμη ευρωπαϊκή που γίνεται όλο και πιο ευρωσκεπτικιστική. Είναι ένα σήμα που δείχνει ότι κινείται και δρά καινοτομή η Ευρώπη, βρίσκει λύσεις για συμπροματικά έσοδα πέρα από επαναλαμβανόμενες διακηρύξεις για λιτότητα που γίνονται και που γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Άρα ε, δίνει η Ευρώπη στον εαυτό της μέσα παρέμβασης, αντί να απλώς να δέχεται παθητικά την κατάσταση. Ναι, σε αυτό το φόρο, σε αυτό το, με αυτό το φόρο η Ευρώπη δείχνει ότι μπορεί να προχωρήσει, ότι δεν χρειάζεται συστηματική προσφυγή στην ομοφωνία όσον αφορά τα θέματα της φορολόγησης. Η φορολόγηση των χρηματοστατικών συναλλαγών δείχνει ότι κάτι είναι εφικτό. Ναι, ε, ε, είναι, έχει, είναι υπερτροφικός τομέας ο χρηματοστητικός. Υπάρχουν κρυμμένοι θησαυροί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις αναγκαίες επενδύσεις, για μια μετάβαση οικονομική και για μια αλλαγή ενεργειακή και οικολογική. Είναι εφικτό με το δρόμο που μας ανοίγει ο φόρος αυτός ναι, είναι μια πρώτη πράξη για, τις, για, τους, για τους ίδιους πόρους, τους δημοσιονομικούς της Ευρώπης. Είναι μια άλλη λογική που μπορεί να ανθίσει για πέρα από την εθνική συμμετοχή υπό τον όρο που ισχύει αυτό που είπε ο συνάδελφος του κόμματος του ΕΛΚ ότι αυτός ο φόρος προστίθεται στις συνεισφορές των κρατών ε, και δεν πάμε σε μηδενικό αποτέλεσμα. Συμφωνούμε απολύτως με την έκθεση της κυρίας Ποδήματα, θα υποστηρίξουμε τις τροπολογίες της και όλος ιδιαίτερος όλες τις τροπολογίες που ευνοούν καλύτερη συλλογή ίσπραξη αυτού του φόρου και κυρίως όλες τις τροπολογίες που καλούν αυτή η φορολόγηση να καλύπτει στο μέγιστο ε, όλα τα μέσα και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Έχουμε κάποια συνεχή ανησυχία όμως όταν συζητούμε τις τροπολογίες θέλουμε αυτή η φορολόγηση, η χρήση αυτού του φόρου να παραμείνει όσο το δυνατόν πιο πιστή ε, στον πρώτο στόχο που έχει, τον αρχικό στόχο του φόρου, δηλαδή να βοηθήσει τις χώρες του Νότου να αναπτυχθούν, να αναπτυχθούν βιώσιμα, να βοηθήσουμε τις χώρες να προστατευθούν από τις συνέπειες της ε, οικονομικής, οικολογικής κρίσης, να βοηθήσουμε εν γέννη να υπερασπιστούν τα, τα παγκόσμια αγαθά, τα δημόσια, τα ύδατα, τα εδάφη, το κλίμα, τα δάση. Ε, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπέσετ. Επόμενος ομιλητής, σαν πολύ Γκοζές. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν δύο ζητήματα σε ό,τι αφορά αυτό τον φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Έχουμε από τη μία το όνειρο και από την άλλη τη σκληρή πραγματικότητα. Το μαγευτικό αυτό όνειρο είναι αυτό το που μας περιέγραψε ο Ζαν Πολ Μπεσέ και με το οποίο και συμφωνώ. Ε, όλα αυτά που είπε ήταν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ενδιαφέροντα και πραγματικά μας παρακινούν. Αλλά αν δει κανεί από κοντά σήμερα τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται κανείς να εφαρμόσει στην πράξη αυτό το φόρο, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές εκπλήξεις. Έχουμε την βασική αρχή, χαμηλή φορολόγηση όλων των συναλλαγών για να έχουμε έναν πόρο, βέβαια πάντοτε ε, με αίσθημα δικαιοσύνης και τα λοιπά. Και είμαι υπέρ όλων αυτών και έχω υπερψηφίσει και τις εκθέσεις της Άννης Ποδηματά χωρίς ε, φόβο και χωρίς πάθος. Αλλά σήμερα βλέπω πραγματικά στην πράξη τι γίνεται. Εκεί το πρόβλημα και Έχουμε και τον ε, Finance Watch, τον ε, οργανισμό αυτό που ενδεχομένως να μην έχει τις ίδιες ιδέες, αλλά με έχει βοηθήσει ε, και στη σκέψη μου και στην επεξεργασία αυτού του θέματος. Βλέποντας λοιπόν από κοντά πώς έχει η κατάσταση, ο τρόπος με τον οποίο έχει οριστεί το παιδί εφαρμογή, βλέπουμε ότι για κάποια χρηματοψηφιακά ιδρύματα αυτά που πληρώνουν τελικά τους φως και όχι ο αν θέλετε, ο επενδυτή, αυτοί, αυτοί οι οργανισμοί τον πληρώνουν και μπορεί μάλιστα να απορροφήσει και το σύνολο των κερδών των τραπεζών αυτών, παραδείγματο χάρη. Έχω ε, στοιχεία, έχω παραδείγματα, μπορώ να σα τα διαθέσω. Και πέραν των αρχών που με βρίσκουν σύμφωνο, όπω είπα, πέραν των στόχων που επίση με βρίσκουν σύμφωνο, πρέπει να έχουμε τη βούληση να δούμε τα πράγματα από κοντά. Γιατί τα νούμερα που βγαίνουν από του υπολογισμού ανθρώπων οι οποίοι εξετάζουν ακριβώ τα πράγματα ω έχουν, καταλήγουν ε, σε μία προσέγγιση πολύ σημαντικότερη σε σχέση με αυτά που μα είπε η Κομισιόν. Θα πει κανεί, ναι, α, μα καλό είναι αυτό γιατί θα έχουμε πιο πολλού πόρου. Μα εδώ δεν πρέπει να αυταπατώμε, θα μιλάμε για πόρου που θα μπορούμε να εκμεταλλευτούμε μετά από 20-30 χρόνια. Και επίση έχουμε ένα πολύ σοβαρό κίνδυνο κατάσταση ή μπορούν να μπουν σε κίνδυνο ιδρύματα τα οποία μόνο λειτουργούν, δεν κάνουν κάτι κακό. Άρα πρέπει να σεβόμαστε τις αρχές σίγουρα και επαναλαμβάνω προσυπογράφω 100% τις αρχές αυτές, αλλά θα πρέπει και η Κομισιόν να κληθεί, να κοιτάξει από πολύ κοντά, πολύ προσεκτικά τι επιπτώσεις θα είχαν κάποιες διατάξεις που ενδέχεται να είναι οδυνηρές και αντιπαραγωγικές και στο οικονομικό επίπεδο και στο επίπεδο των φορολογικών εσόδων. Διότι αν η φορολογική βάση εξαφανιστεί, θα υπάρχει μεν φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, αλλά δεν θα έχει την επίπτωση που θέλουμε. Σήμερα λοιπόν υπάρχει αυτό ο κίνδυνο σε κάποιου τομεί και για κάποιε συγκεκριμένε περιπτώσει να ε, βλέπουμε αυτό το κίνδυνο να υπάρχει ο κίνδυνο εξαφάνιση αυτή τη βάση τη φορολογική. Δεν είμαι πολύ British, αλλά επειδή λέμε συχνά αυτή την έκφραση ότι ο διάβολος στις λεπτομέρειες κρύβεται, εγώ θα έλεγα ότι για να πάμε στον παράδεισο πρέπει να σκοτώσουμε τον διάβολο στην προκειμένη περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ κύριος Γκίκολτ τώρα. Um, first I, Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ ότι πλέον ο διάβολος ε, κρύβεται στις λεπτομέρειες και η λεπτομέρεια έχει σημασία Είτε ο φόρος αυτός τελικά στραφτεί με επιτυχία, είτε όπως και άλλοι φόροι τελικά καταλήξει στο καλάθι των ε, προσπαθειών με καλές προθέσεις. Γιατί αν τελικά καταλήξουμε εκεί, ε, θα έχουμε αποτύχει. Γιατί η ιδέα ήταν να υπάρχει ένας καθολικός φόρος για το δημόσιο χρέος, και για να υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο μια εξισορρόπηση. Αν προχωρήσει τώρα ε, μια ομάδα μόνο κρατών με το φόρο αυτό, θα πρέπει να ε, είναι σωστή η εφαρμογή του. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι ευρεία η βάση για να αποφευχθεί οποιαδήποτε δυνατότητα αποφυγής του φόρου. Στο παρελθόν το Κοινοβούλιο ε, σωστά έκανε και πρότεινε να προσθεθούν μέτρα για την ε, πρόληψη της φοροαποφυγής στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ιδάλλως αν καταλήξουμε να κάνουμε κάτι παρόμοιο με τη Σουηδία, τελικά θα έχουμε, πράξει, θα έχουμε διαπράξει ένα τεράστιο σφάλμα. Γιατί φυσικά Εξακολουθούμε να θέλουμε ένα καθολικό φόρο. Καθολικό φόρο θα πετύχουμε μόνο αν μπουν όλες οι χώρες και θα μπουν όλες οι χώρες μόνο εάν σταθεί με επιτυχία ο μηχανισμός αυτός και αν τα χρήματα αυτά χρησιμοποιούνται για στόχους που θα βρίσκουν συμφωνές όλες τις χώρες. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να διαπραγματευτούμε και με άλλες χώρες σε διεθνές επίπεδο την επιβολή ενός τέτοιου φόρου. Όπως ξέρετε, η ο χρηματοπιστωτικός κλάδος είναι καινοτομικός, παρά το γεγονός ότι δεν ξέρουμε αν αυτή η καινοτομία εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον ή όχι, αλλά όντω χαρακτηρίζεται από καινοτομία. Άρα καλό θα ήταν να υπάρχει μια μόνιμη επιτροπή που θα παρακολουθεί τι γίνεται με την επιβολή του φόρου αυτού και αυτό κινείται προς την κατεύθυνση του Ζαν Πολ. Φυσικά ένας λόγος είναι να μειωθεί η φορολογική βάση. Θα ήταν αντιφατικό να λέγαμε ότι έχουμε φόρο επί των χρηματοπιστωτικών ε, ε, συναλλαγών και μετά ε, λέμε ότι διαβρώνεται η φορολογική βάση. Όχι, αυτός είναι ένας βασικός στόχος. Αλλά τι δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε ο κλάδος, ο οποίος έχει διαβρωθεί στην Ευρώπη, να ανακύψει κάπου αλλού στον κόσμο από τους ίδιους φορείς. Αυτό προσπαθούμε να αποφύγουμε. Θέλουμε να περιορίσουμε την κοντοφθαλμία αλλά θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί σε θέματα φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Και φυσικά, υπό την όνεια αυτή, κανείς δεν ξέρει πώς πραγματικά θα αντιδράσουν οι αγορές. ηρεώσουμε την πρόταση αυτή, η οποία την χάνει διαπραγμάτευση ε, υπό τη διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας, αλλά επιμένουμε να παραμείνει ανοιχτό σύστημα αυτή η διαπραγμάτευση, δηλαδή να μπορεί να προσαρμόζονται σε όλες τις χρηματοπιστωτικές καινοτομίε που είμαστε βέβαιοι ότι θα ανακύψουν. Και γι' αυτό λοιπόν σε ό,τι αφορά τις εξαιρεσει που έχουν συζητηθεί και στο παρελθόν στο Κοινοβούλιο, όπως και τα συνταξιδοτικά ταμεία για παράδειγμα. Θεωρώ ότι όλα αυτά τελικά θα υπονομεύσουν την αποτελεσματικότητα τον, ε, του φόρου θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας χάμηλος συντελεστής και να ισχύει για όλες τις συναλλαγές με πολύ πολύ περιορισμένες εξαιρέσεις όπως προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Σε αυτό το πνεύμα λοιπόν θα πρέπει να συνεχίσουμε και να προσέξουμε ιδιαίτερα προκειμένου τα συμμετέχοντα να έχουν την ευχέρεια να προσαρμόζονται σε οποιαδήποτε νέα μορφή φοροαποφυγής και σε οποιαδήποτε νέα κοινοτομία του κλάδου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γκίγκολτ. Αν δεν ζητάει κανείς άλλο το λόγο, λέει ο πρόεδρος, θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον κύριο Μπέκμαν. Okay, thank you, Chairman, and thank... Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Ποδηματά για την παρουσίαση αυτής της έκθεσης που φυσικά χαιρετίζουμε πολύ από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί στηρίζει πλήρω τη θέση της Κομισιόν, καταρχήν τουλάχιστον, σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα, το φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Σε κάποιε ε, βέβαια, περιπτώσεις ενδεχομένως πηγαίνει λίγο πιο μακριά από την πρόταση τη Κομισιόν, ιδίω ό,τι αφορά τι προθέσεις για ενίσχυση τις διατάξεις ε, κατά της αποφυγής. Θέλει επίσης να υπάρξει μεγαλύτερη λεπτομέρεια και μεγαλύτερη εναρμόνιση ε, στη συλλογή στοιχείων και επίσης περιλαμβάνει και κάποιες πολιτικές δηλώσεις που κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπερβαίνουν λίγο ε, αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε ότι θα ήταν απαραίτητο σε ένα τέτοιο νομικό κείμενο. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της μέγιστης εναρμόνισης, γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθούσε πάντοτε στον τομέα της έμεσης φορολόγησης την προσέγγιση της όσο το δυνατόν περισσότερης εναρμόνιση, αλλά όσο αυτό είναι αναγκαίο για να λειτουργήσει η εσωτερική αγορά. Στον τομέα της φορολόγηση, θέλουμε να προτείνουμε ελάχιστου συντελεστέ, αλλά να αφήσουμε τα κράτη-μέλη να αποκλίνουν ενδεχομένω ή να υιοθετήσουν υψηλότερα ποσοστά υψηλότερου συντελεστέ. Γνωρίζουμε όμω ότι ιδίω ό,τι αφορά κινητέ βολοκέ βάσει, όπω είναι τα παράγωγα για παράδειγμα, εκεί ο ελάχιστο συντελεστή θα μπορούσε να είναι ο συντελεστή που θα εφαρμόζεται στι χώρε. Επίση, ε, σε ό,τι αφορά ε, την ενίσχυση των διατάξεων κατά της αποφυγής, ναι, να ενισχυθούν, συμφωνούμε. Ωστόσο, πάντοτε πρέπει να έχουμε υπόψη μας την ανάγκη για εξέβρεση μιας καλής ισορροπίας. Αφενός δηλαδή να ενισχύσουμε το σκέλος της ε, αντιαποφυγής, από την άλλη όμως να εμείνουμε στο πλαίσιο ε, των, ε, της νομοθεσίας για την εμισφορολογία και νομίζω ότι ίσως προκύψουν κάποια προβλήματα. Με βάση την προτινόμενη έκθεση φοβούμεθα ότι αν ακολουθήσουμε το μονοπάτι που προτείνει εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ίσως να είναι πολύ αδύναμος ο γεωγραφικός σύνδεσμος ε, για, τη, ε, για το φόρο, διότι πολλές φορές κατηγορούμαστε ότι προωθούμε τον εξοεδαφικό χαρακτήρα. Εδώ όμως είμαστε αισιόδοξοι και επιπισμένοι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση, γιατί πάντοτε ελέγχουμε κατά πόσο υπάρχει σύνδεσμος, υπάρχει σχέση μεταξύ της οικονομικής ουσίας μιας συναλλαγής και του, της επικράτησης ενός κράτους μέλους. με την ε, γραμμή όμως που ακολουθεί ή που προτείνει η έκθεση, ίσως ισως παψει να υπάρχει επαρκή σύνδεσμο σε σχέση μεταξύ της συναλλαγής και της επικράτειας του κράτους μέλους. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, εφαρμογή, τη συλλογή κτλ. Ε, η εισπράξη μάλλον αυτού του φόρου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί ότι χρειάζεται εδώ εναρμόνιση, πολύ εναρμόνιση και για να έχουμε μια καλή σχέση κόστος-οφέλους, γιατί μιλάμε για κινητή, ε, ευέλικτη φορολογική βάση. Πρέπει να υπάρχουν λοιπόν ε, παρόμοιες διατάξεις και στο αφορά τις υποχρεώσεις των κρατών μέλων. Το θέμα είναι όμως, πρέπει εδώ να γίνει συγκεκριμένη πρόταση και να το αφήσουμε στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν για την συντονισμένη προσέγγιση που θα θέλουν να ακολουθήσουν. Είναι σαφές ότι η Κομισιόν, σε περίπτωση που θέλουν τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε μεγαλύτερη εναρμόνιση, συμφωνεί ότι ίσως είναι απαραίτητο για να υπάρχει βέλτιστη σχέση ε, κόστους-οφέλους, αλλά και αν θέλουν οι χωρίς μέλη να προσεγγίσουν εταίρους από τρίτα κράτη. Ίσως ήταν καλό να υπάρχει μια ομαδική προσέγγιση από πλευράς κρατών μελών προς αυτές τις δικαιοδοσίες και προς αυτές τις υποδόμες τρίτων κρατών. Και έρχομαι στο τελευταίο μου σχόλιο. Το αίτημα ορισμένων βουλευτών να υπάρξουν κάποιες παρεκκλήσεις, εξαιρέσεις, ειδική μεταχείριση σε συγκεκριμένα θέματα. Θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι αν αυξάνουμε τον αριθμό των εξαιρέσεων και των αποκλήσεων, θα είναι πολύ δύσκολο ε, να εισπράτεται αποτελεσματικά και οικονομικά αυτός ο φόρος. Υπάρχουν κάποια επιχειρήματα κάποιοι που ζητούν αυτές τις εξαιρέσεις και πρέπει να τα μελετήσουμε και αυτά, αλλά θα πρέπει να δούμε και ποιο θα ήταν το σωρευτικό αποτέλεσμα των προνομίων. Σκεφτείτε τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η επένδυση σε ε, συνταξιοδοτικά ταμεία ήδη ε, έχει, ε, η επένδυση αυτή έχει προτιμησιακή μεταχείριση σε σχέση με άλλες μορφές αποταμίες, ταμείες για την σύνταξη, για τη συνταξιοδότηση και αν δώσουμε και εδώ άλλο ένα κίνητρο, ίσως το παρακάνουμε. Πάντα λοιπόν θα πρέπει να θέτουμε το ερώτημα to tax or not to tax. Να φορολογήσουμε ή να μην φορολογήσουμε. Το θέμα είναι να μην επηρεαστεί η αρνητικά λειτουργία των αγορών. Και εδώ αναφέρομαι στο αίτημα της διαχείρισης του δημοσίου χρέους. Κατά εμάς δεν είναι θέμα να φορολογηθεί όχι δευτερογενής ε, αγορά. Το θέμα είναι να φορολογηθεί με τρόπο τέτοιο που να βοηθήσει τη λειτουργία αυτών των δευτερογενών αγορών. Ο κύριος Γκίκολτ είπε, νομίζω, ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δείξουν ότι λειτουργεί πρώτα πρέπει να έχουμε σωστά τη μελέτη, το σχεδιασμό και μετά να δούμε τη φάση της ε, ίσπραξης του φόρου, της πρακτικής εφαρμογής δηλαδή αυτού του συστήματος. Συμμεφετήρες καταρχάς θα πρέπει να είναι αυτή η ομάδα των 11 και θα ακολουθηθεί ο παραδοσιακός τρόπος ευρωπαϊκής ολοκληρωσής όπως ξεκίνησε στη δεκαετία του 50. Είχαμε ξημέλη, και μόνο για την αγορά του άνθρακα και του χάλιβα και τώρα έχουμε φτάσει σε 27, ε, σύντομα 28 και το ίδιο ελπίζουμε να συμβεί και με το φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Δηλαδή άπαξ και εφαρμοστεί από τα 11 κράτη και φανεί από αυτά ότι παράγεται παράγονται έσοδα χωρίς να ε, επηρεάζει τα αρνητικά λειτουργία των αγορών, θα ακολουθήσουν και άλλα κράτη-μέλη και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός. Ίσως δηλαδή και άλλοι αποφασίσουν να εισαγάγουν αυτό το φόρο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο εν τέλει στην εισηγήτρια. Κυρία Ποδηματά, έχετε το λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, Ραμόν. ξεκινώντα από το τελευταίο σημείο που έθεσε ο κύριος Μπέργκμαν, αλλά που αναφέρθηκε και από κάποιου από τους προλαλήσαντες και τους κοιόδης εισηγητές. Σίγουρα, αναμφισβήτητα, ένας από τους στρατηγικούς μας στόχους μέσω της έγκρισης της διευρυμένης συνεργασίας για την εφαρμογή του φόρους χρηματοπιστωτικών συναλλαγών από 11 κράτη-μέλη σε μια πρώτη φάση είναι κάτι που σημαίνει ότι θέλουμε να δείξουμε ότι αυτός ο φόρος είναι κάτι εφικτό, αποδοτικό, αποτελεσματικό ούτως ώστε να ενθαρρυνθούν άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να συμμετάσχουν σε αυτή τη λέσχη τι ούτω τρόπος θα αναζαγωνηθεί η εκστρατεία μας και η προσπάθειά μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κινηθούμε προς ε, παγκόσμιο φόρο, γενικό φόρο φορολόγησης ε, χρηματοστικών συναλλαγών, διότι όπως αναφέρομαι σε σχέδιο εκθέσεως, σε μία τροπολογία μου, αυτός ο φόρος χρηματοδοτικών συναλλαγών θα παράγει τα πλήρη αποτελέσματα τα οποία μπορεί όταν εφαρμοστεί σφαιρικά, γενικά, παντού. Είναι σαφέστατο αυτό. Και είναι κοινή άποψη του Κοινοβουλίου. Αν θέλετε να ενισχύσουμε ε, περαιτέρω αυτή τη δέσμευση και αυτό το στόχο, εγώ είμαι απόλυτα θετική. Και κάτι άλλο, ένα άλλο σημείο το οποίο την χάνει ευρεία συνενέσεως, τουλάχιστον μεταξύ των σκιωδών εισηγητών, και μακάρι να είναι σημάδι ευρυτέρων συνενέσεων εντός των πολιτικών ομάδων αυτό, αφορά τη διαχείριση των πόρων. Και όλος ιδιαίτερος τη σχέση με τους ιδίους πόρους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η πρότασή σας να διευρύνουμε περαιτέρω να αυξήσουμε τις αναφορές τις σχετικές ε, με βρίσκει σύμφωνη και δεύτερον η πόρη από το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σαν μη πόρη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σαν, ίδιοι, σαν ίδιοι πόροι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν θέλουμε να αντικαταστήσουν τις συνεισφορές των κρατών μελών αλλά θέλουμε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτός είναι ένας στόχος που ενστερνίζομαι και εγώ και η ομάδα μου. Ελπίζω και εύχομαι να υπάρξει συνένεση στο Κοινοβούλιο και εντό των μεγαλύτερων πολιτικών ομάδων σχετικά με αυτό, τούτου λεχθέντος, επαναλαμβάνω κάτι που και ο κύριος Μπέρκμαν ε, ανέφερε. Είναι σημαντικό και σημαντικό σαν πολιτική δήλωση δεν μπορεί να επηρεάσει όμως το νομικό τμήμα του σχεδίου οδηγίας. Αυτού του είδους οι αναφορές είναι σημαντικές πολιτικός πως, το υπογραμμίζω αυτό εκ νέου, όμως μπορούν να αποτελέσουν ένα τμήμα μόνο των αναφορών που συμπεριλαμβάνουμε στις αιτιολογικές σκέψεις. Έρχομαι τώρα σε πιο συγκεκριμένες προτάσεις και σχόλια που εκφράσατε. Η θέση μου σχετικά τις ενδεχόμενες εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής του φόρου καταρχήν είναι αρνητική και νομίζω ότι εξήγησα το λόγο. Νομίζω ότι όσο πιο πολύ δημιουργούμε περιθώρια εξαιρέσεων, τόσο δημιουργούμε περιθώρια για μειωμένη απόδοση και αποτελεσματικότητα στον αφορά την εφαρμογή του φόρου. Αυξάνουμε τις δυνατότητες φόρο και φόρο οπότε χωρίς να είμαι δογματική, καταρχήν πιστεύω ότι θα πρέπει να αποφύγουμε τις εξαιρεσει και αυτό ταιριάζει με αυτό που συνεφώνησαν καταρχήν τα κράτη-μέλη που το ζήτησαν με επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σεβασμό της αρχικής πρότασης, δηλαδή θέλουμε την ευρύτερη δυνατή κάλυψη όσον αφορά το φόρο αυτό. Για τα δύο συγκεκριμένα θέματα που εθίγησαν και τις ερωτήσεις, πρώτα απ' όλα το θέμα των συνταξιδοτικών ταμείων. Αυτό είναι κάτι που έχει συζητηθεί στη, σε προηγούμενη έκθεση. Είναι κατανοητό ότι είναι θέμα ανησυχίας για κάποιους από εσά, κάποιους από εμά, να επενθυμίσω εκ νέου κάτι. Μία κοινή θέση που έχουμε καταρχήν ότι αυτά τα ταμεία θα πρέπει να ακολουθήσουν συντηρητική, μάλλον συντηρητική επενδυτική πολιτική. Και εν γέννη θα συμφωνείτε ότι τα συντεξιδοτικά ταμεία δεν καλούνται να κερδοσκοπούν ή να έχουν τεράστιες δαπάνες συναλλαγών. Αυτό συνάδει με το βασικό σκοπό που έχει ένα συνταξιωτικό ταμείο που μη λησμονούμε είναι να καταβάλει σύνταξη μετά από 20 ή 30 χρόνια οικονομιών και αποταμιεύσεων. Για τη δευτερογενή αγορά τίτλων μετοχών που έθεσε ο Ραμόν σε προηγούμενη συνεδρίαση, αλλά τον έφερε και σήμερα. Ήθελα να επιθυμίσω κάτι. Πρόσφατη μελέτη του City του Λονδίνου όσον αφορά την επίδραση του φόρου είναι ότι είναι 11,6% όσον αφορά τις συναλλαγές και υποθέτει ότι κάθε συναλλαγή τίτλου θα δίνει 5 φορολογήσιμα γεγονότα. Αυτή είναι μια υπόθεση εσφαλμένη, διότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξαιρεί στη διαμεσολάβηση όταν ένα χρηματοδοτιστικός, ένα χρηματοδοτιστικός φορέας εν ονόματι και για λογαριασμό άλλου χρηματοδοτικού φορέα. Και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την αξιολόγηση συνεπιών που έκανε, ο αντίκτυπος, η συνέπεια, σας την πεθυμίζω, στη δανειοδότηση κυβέρνησης είναι στο 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ και το εισόδημα είναι 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ε, είναι θετικό αποτέλεσμα για, τα, για τους υπολογισμούς των κρατών μελών. Σίγουρα όμως θα πρέπει να συζητήσουμε περαιτέρω το θέμα και να το εξετάσουμε ενδελεχέστερα. Σχετικά με την πρόταση που κάνατε κάποιοι να αντικαταστήσουμε τα ελάχιστα ποσοστά που συμπεριλαμβάνονται στην πρώτη Ευρωπαϊκή Ενώσεω με ενιαία ποσοστά Θέλουμε να κρατήσουμε τα ελάχιστα ποσοστά ως προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό πρέπει να το κάνουμε κατά πρώτον, διότι οι αγορές θα αντιδράσουν σίγουρα με διαφορετικό τρόπο και όπως είπατε κάποια από εσά, δεν γνωρίζουμε ακριβώς το πώς θα αντιδράσουν οι αγορές. Συνεπώς πιστεύω ότι αν κινηθούμε βάσει της παρούσης προτάσεως και καταρτήσουμε ε, ε, ελάχιστα ποσοστά και διαφοροποιημένα ποσοστά στις διάφορες αγορές, ε, είναι η καλύτερη προσέγγιση και πιστεύω ότι εάν η πρότασή μας εγκριθεί Δηλαδή να δημιουργηθεί μια ομάδα για το φόρο χρηματοσωτικών συναλλαγών που θα πρέπει τακτικά να αξιολογεί την πορεία των πραγμάτων, τότε θα μπορούσαμε να λάβουμε την εντολή να αξιολογήσουμε το θέμα, δηλαδή να δούμε κατά πόσο αυτή η διαδικασία, αυτή η ευελιξία για τα κράτη-μέλη που θα μπορούν να αλλάζουν τα ποσοστά, να τα αυξάνουν, αν είναι η καλύτερη λύση ή αν πρέπει να προχωρήσουμε σε μια δεύτερη φάση. Στην πρώτη αναθεώρηση, επί τη ευκαιρία της πρώτης αναθεωρήσεως της οδηγίας για το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και φτάσουμε σε εναρμονισμένο φόρο εναρμονισμένο ποσοστό σε αυτά και ελπίζω να μην ξέχασα κάτι σημαντικό μέχρι τώρα. Σα ευχαριστώ για μία ακόμη φορά για τα σχόλιά σας, για τις προτάσεις σας και εν γέννη για τη συνεργασία σας. Κυρίως ευχαριστώ τους σκιώδεις εισηγητές και προσβλέπω στη συνέχιση αυτής της καρποφόρας συνεργασίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ραμόν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ποδήματα. Να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία υποβολή τροπολογιών είναι 23 Απριλίου η συζήτηση των τροπολογιών θα λάβει χώρα στις 27 Μαΐου, η ψηφοφορία στην Επιτροπή 28 Μαΐου και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια αναμένεται να λάβει χώρα τον Ιούλιο. Τούτων λεχθέντων προχωρούμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Θα συζητήσουμε τις τροπολογίες της εκθέσεως της κυρίας Γκάλ Πέλες για την ετήσια έκθεση για φορολόγηση Πώ να απελευθερώσουμε το δυναμικό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω για την οικονομική ανάπτυξη. Δίνω το λόγο λοιπόν στην κυρία Γκάλ Πέλε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Επιτρέψτε μου καταρχάς ε, να σας ευχαριστήσω για τις ε, πολλές ε, τροπολογίες. 144 στον αριθμό. και θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατατάσσονται σε κάποιες μεγάλες ε, κατηγορίες. Ο πράσινος φόρος, ε, φοροδιαφαγή, φοροαποφυγή. Πριν ε, τις πασχαλινές διακοπές, καταφέραμε με τους σκιώδεις εισηγητές να ορίσουμε το διάγραμμα, αν θέλετε, των ε, συμβιβαστικών προτάσεων. Και έχω ήδη λάβει απαντήσεις για τις συμβιβαστικές προτάσεις αυτές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σκοπός της εργασίας μου ήταν στην ε, τρέχουσα δύσκολη χρηματοπιστωτική και οικονομική συγκυρία τα φορολογικά συστήματα να εξυπηρετήσουν τον απότερο στόχο της οικονομικής ανάπτυξης και ανάκαμψης ως εκ τούτου θεωρώ ότι στόχος είναι να τονίσουμε την στρατηγική της Ευρώπης 2020 και τα διάφορα φορολογικά μέτρα τα οποία θα πρέπει να εξυπηρετούν ακριβώς αυτό το σκοπό. Ωστόσο, μπορώ να αποδεχτώ, να και παρακαλώ και τους συναδέλφους να το αποδεχτούν αυτό, ότι οι οικονομικές και αφορολογικές πολιτικές στα διάφορα κράτη είναι διαφορετικές. Ε, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις απαντήσεις ε, που δίνονται στην κρίση, αλλά και την ε, κατάσταση που επικρατεί στην κάθε χώρα και αυτό αναλόγως επηρεάζει με διαφορετικό τρόπο και τις φορολογικές πολιτικές στα, κάθε κρατη, στα μελη Φυσικά μιλάω και για θέματα ηθικής διαντολογίας σε ό,τι αφορά την ίσπραξη των φόρων, αλλά και για θέματα ε, διαφάνειας. ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το Φισκάλις αναφέρω ότι θα πρέπει να λειτουργούν σωστά. Τονίζω επίσης την έκθεσή μου ότι σε ό,τι αφορά τους εταιρικούς φόρους, το πρόβλημα των αυτοαποσχολουμένων θα πρέπει να ε, το προσέξουμε ιδιαίτερα. Τώρα σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ, τόνισα ότι καλωσορίζουμε και θα καλωσορίζαμε ιδιαίτερως ένα ενιαίο συντελεστή φορολογίας, γιατί όταν ε, αν απελευθερωθούν, για παράδειγμα, θέματα πολιτισμού ή τα τρόφιμα από το φόρο αυτό. Αυτό θα επηρεάσει βαθύτατα σε βραχυπρόθεσμο όμως πλαίσιο, ο καταναλωτής δεν θα το νιώσει αυτό, γιατί η μείωση του ΦΠΑ αποτελεί ένα buffer, αν θέλετε, ένα ενδιάμεσο επίπεδο και ίσως ε, με τον χαμηλό φορολογικό συντελεστή σε θέματα πολιτισμού ε, θα δοθεί έτσι βραχυπρόθεσμα, ένα κίνητρο. Μακροπρόθεσμα όμως δεν μπορεί να είναι χρήσιμο κάτι τέτοιο. Αυτό αποτελεί προσωπική μου άποψη. Ευχαριστώ όμως να ακούσω και την άποψη των συναδέλφων. Την άλλη εβδομάδα θα συναντηθούμε με τους σκιώδεις συζητητέ. Τώρα σε ό,τι αφορά τη Στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση 2020. Τόνισα ότι θα ήταν απαραίτητο να εισαχθεί μια φορολογική πολιτική η οποία θα ενισχύει την παραγωγικότητα και την απασχολησιμότητα. προκειμένου να μην διακυβεύονται θέσεις εργασίας. Και θεωρώ ότι αυτό θα αυξήσει και την αποδοχή από τους κοινωνικούς εταίρους. Άλλα δύο θέματα θα ήθελα να αναφέρω, τα οποία θεωρώ ότι είναι σημαντικά. Καταρχάς, το ζήτημα του φόρου για, του περιβαλλοντικού φόρου και το θέμα της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής κάνω την Ο συνάδελφος έχει ε, μία έκθεση με παρόμοιο θέμα, γι' αυτό λοιπόν θέλησα να αποφύγω ε, επαναδιατυπώσεις και αλληλεπικαλύψεις στη δική μου έκθεση. Γι' αυτό, σε ό,τι αφορά τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποφυγή ε, διπλής φορολόγηση την αποφύγη των φορολογικών οάσεων. Ε, τα ανέφερα αυτά και σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται και οι τροπολογίες μου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πράσινη φορολογική πολιτική, δεν τόνισα τόσο πολύ τους πράσινους φόρους, όσο ιδιαίτερος τους φόρους εκείνους που θα διευκολύνουν μία τροποποίηση της φορολογικής πολιτικής. Θεωρώ ότι αυτές, αυτή είναι πιο σωστή. Αυτά τα μέτρα είναι πιο σωστά. Στις 20 συμβιβαστικέ προτάσεις ακολούθησα αυτή τη γραμμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεργασία σας και προσβλέπω στην συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Τώρα εξ ονόματων σοσιαλιστών, ο κύριος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχά θέλω να ευχαριστήσω την συγκεκριτή για την πολύ καλή μέχρι τώρα συνεργασία μα. Ήταν πάρα πολύ θετικέ οι πρώτε συμβαστικέ προτάσει ε, και νομίζω ότι η συζήτηση πηγαίνει προ τη σωστή κατεύθυνση. Η έκθεση αυτή είναι σημαντική για αρκετού λόγου. Ε, η πιο επίγουσα ε, πτυχή είναι ότι θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχει σαφής διασύνδεση μεταξύ φορολογικής πολιτικής και ανάπτυξης. Και αυτό πρέπει να το τονίζουμε, να το τονίζουμε διαρκώς. Είναι από φασιστική σημασία να έχουμε ένα καλό ε, ισορροπημένο και καλώς λειτουργούν ε, φορολογικό σύστημα για να πετύχουμε και την ανάπτυξη που είναι απαραίτητη. Αλλά υπάρχει ένα ερωτηματικό σε ό,τι αφορά αυτό το φορολογικό ε, φίδι ε, το οποίο προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και για το πώς θα συντονίσουμε όλα τα συστήματα. Χρειάζονται λοιπόν περιττέρω διευκρινήσεις. Γιατί αν απλά αντιγράψουμε ε, το νομισματικό φίδι που ήταν τα πρώτα στάδια της συνεργασίας πριν από τη μετάβαση στο ευρώ. Αυτό, κατά την άποψή μου, θα σημάνει ε, πολύ μεγάλη φορολογική εναρμόνιση με ανώτερα και εκατώτερα όρια και έχω κάποιες αμφιβολίες σε σχέση με την προσέγγιση αυτή. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ήδη κάποια εναρμόνιση στα φορολογικά επίπεδα, γιατί έχουμε τεχνικούς κανόνες και κατώτατα επίπεδα. Αλλά αυτό είναι καλό. Αλλά αν θέλουμε να βάλουμε μέγιστα όρια, δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν ευκταίο. Τουλάχιστον στην παρούσα χρονική στιγμή. Χωρίς περαιτέρω εναρμόνιση, νομίζω ότι παρόλα αυτά μπορούμε να βελτιώσουμε τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών και αυτό θα ήταν ένα θετικό βήμα. Νομίζω ότι θα είναι και ένα βήμα σημαντικό προς τη σωστή κατεύθυνση. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να αποφύγουμε τον όρο φορολογικό φίδι, tax snake. Γιατί μπορεί κάποιοι να κάνουν τους λάθος συνειρμούς ε, με ένα τέτοιο όρο και πρέπει να το συζητήσουμε νομίζω σε μεγαλύτερο βάθος. Όσο προχωρούν οι εργασίες μας ε, θα ε, αναπτύσσω και τις απόψεις μου, αλλά τώρα θέλω να αναφερθώ σε τέσσερα σημεία. Πρώτον, πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας κατά της φοροαπάτης και της φοροδιαφυγής. Αυτό θα είναι ένα σημείο κλειδί για να δημιουργηθούν ε, οι απαραίτητες περιποθέσεις για βιώσιμη και μακροχρόνια ανάπτυξη, γιατί θα ενισχυθούν τα δημόσια οικονομικά θα ε, ευνοηθεί ο θεμητός ανταγωνισμός και αυτό θα αυξήσει και τον απτυξιακό δυναμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επόμενο σημείο. Πρέπει η ανάπτυξη να ενισχυθεί με την άρση φορολογικών εμποδίων στην εσωτερική αγορά. Η οδηγία για τον ΦΠΑ θα πρέπει να οδηγήσει σε βελτιώσει στον τομέα αυτό. ένα ενοποιημένο κείμενο θα μπορούσε και αυτό να βελτιώσει και τη συνεργασία ή η βελτίωση ε, της, ε, υπουργικής, ε, της υπουργικής συνεργασίας και με τις φορολογικές αρχές. Τρίτον, πρέπει να δούμε τις κοινωνικές πτυχές που πρέπει να συμπεριλάβουμε και στην έκθεση αυτή. Δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε φορολογικές δομές που θα αυξήσουν το χάσμα στην κοινωνία. Το χάσμα πλουσίων και φτωχών δεν είναι από μόνο του αρνητικό, αλλά επηρεάζει αρνητικά και την ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνει, το, αυξάνει τους φόρους κατανάλωσης, που όμως τελικά ε, επηρεάζουν περισσότερο τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα που επομίζονται ένα μεγάλο μέρος έτσι του φορολογικού φορτίου και δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό. Περιβαλλοντικός φόρος, πράσινος φόρος είναι σημαντική φόρη για να δημιουργηθεί βάση για την ανάπτυξη. Η τάση όμως στην Ένωση είναι να συρρυκνούται αυτός ο πράσινος φόρος και νομίζω ότι αυτό είναι πρόβλημα. Θα ήταν πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για την ανάπτυξη αν οι πράσινοι φόροι ήταν, ε, είχαν μια μεγαλύτερη αναλογία, ήταν ένα μεγα, είχαν ένα μεγαλύτερο μερίδιο στο φορολογικό σύστημα. Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε έτσι και μια ομαλή μετάβαση προς μια πράσινη οικονομία και ένα πρώτο βήμα γι' αυτό θα ήταν η αναθεώρηση και η ενίσχυση της ε, οδηγίας για την ενέργεια. Αυτά είναι τα τέσσερα σημεία μου και αν δουλέυσουμε πάνω σε αυτά νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε καλούς συμβιβασμούς. Όπως είπα, μέχρι τώρα η διαδικασία ήταν πολύ επικοδομητική, δημιουργική και νομίζω ότι είμαστε σε καλή θέση για να συνεργαστούμε και να εκπονήσουμε εξαιρετική έκθεση. Ο πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κύριε Λούτβιξτ. Κύριος Τρεμόσα θα πάρει τώρα το λόγο, μέρος τη Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά που έκανε. Διαβάζοντας τις συμβαστικές Έχω την εντύπωση ότι έχει γίνει σεβαστό το πνεύμα της αρχικής ε, εκθέσεως, οπότε δεν έχω πολύ από αυτού. Όμως, έχω κάποια προβλήματα με την έννοια αυτού του φορολογικού όφεως, διότι πιστεύω ότι αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη είναι να μην έχει μια διαδικασία φορολογικής εναρμόνισης. Ας δούμε τι γίνεται στη ΣΥΠΑ για να μπορούμε να κάνουμε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δούμε και να συγκρίνουμε βέλτιστες πρακτικές. Και είπα έχουν νομισματική πολιτική. Όμως υπάρχει φορολογική ανεξαρτησία για, τα, για τις 50 πολιτείες να αυξήσουν, να μειώσουν φόρους, να καταργήσουν φόρους. Και είναι ένα μοντέλο φορολογικού ανταγωνισμού που κάνει όλη την οικονομία αποδοτική και υπάρχει τεκμηρίωση οικονομική που δείχνει τις διαφοροποιημένες συνέπειες μιας ενιαίας νομισματικής πολιτικής σε διάφορες επικράτειες. Διότι η οικονομική δομή των διαφόρων πολιτιών διαφέρει. Οπότε η φορολογική πολιτική είναι ένα εργαλείο ε, των πολιτιών, των 50 πολιτιών και των ΗΠΑ να μειώσουν τον αντίκτυπο που έχει αύξηση μείωση του, ε, του ποσοστού και του επιτοκίου σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι πολύ πιο ανταγωνιστική η οικονομία από την ευρωπαϊκή, διότι αυτό που εναρμονίζεται στη ΣΥΠΑ είναι η αγορά εργασίας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πολλές διαφορές όσον αφορά τις αγορές εργασίας, διαφορές μεταξύ σκανδιναβικών χωρών και νοτίων χωρών και αυτό δημιουργεί αποκλήσει και διαφορέ, οικονομικέ, μακροοικονομικέ διαφορέ. Πρέπει να δούμε τις διαφορές ε, και στα επίπεδα της ανεργίας. Αυτή είναι η προσέγγιση που πρέπει να ακολουθήσουμε. Όχι με εναρμόνιση των φόρων, να κινηθούμε, αλλά με παραγωγικούς παράγοντες, όπως οι αγορές και η εναρμόνιση της αγοράς κεφαλαίων και της αγοράς εργασίας. Γι' αυτό προσωπικά εγώ είμαι κατά της στρατηγικής αυτής που κάποιοι ευρωβουλευτές προασπίζουν δηλαδή να προχωρήσουμε προς φορολογική εναρμόνιση. Και τελικά αυτό που αφορά και τις τροπολογίες μου. Έστειλα χθε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα σε και στους σκιώδεις εισηγητές και στους διαφόρους συμβούλους προσπαθώντας να βελτιώσω το συμβιβασμό που, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται το όνομά μου. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε σε αυτού του είδους αιτήσει εκθέσεις περί φορολογίας, ότι σε κάποια κράτη-μέλη, περιφέρειες και τοπικές αυτοδιοίκησεις έχουν εξουσίες εισπραξης φόρων καμιά φορά. Γι' αυτό καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το λάβει αυτό υπόψη. Όταν ετοιμάζει προτάσεις να το λάβει υπόψη ότι κάποιες περιφέρειες στην Ευρώπη έχουν ε, μερικές ή πλήρεις ε, δυνατότητες εισπράξης φόρων όπως στη Γερμανία, στην Ισπανία σε δύο από τις 17 περιοχές ισχύει. Οι δύο από 17 περιφέρειες στην Ισπανία έχουν πολύ χαμηλότερα επίπεδα ανεργίας και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Η, η Ναβάρα και η χώρα των Βάσκων, η περιοχή των Βάσκων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και για πολλές άλλες περιφέρειες Όπω στην Καταλωνία, είμαι βουλευτή από την Καταλωνία, είναι πολύ καλή πρακτική. Θα πρέπει να, να επεκτείνουμε αυτή την ε, πολιτική για να βελτιώσουμε τα οικονομικά αποτελέσματα. Γι' αυτό στην τροπολογία 1α, που αφορά την τροπολογία μου 42, θα ήθελα να αντικατοπτρίζεται αυτή η προσέγγιση στη συμβιβαστική τροπολογία. Η ΔΕΜΗ θα αποσύρω το όνομά μου από τη συμβαστική. Όσον αφορά τη συμβαστική, που αφορά την παράγραφο 8 νέα, Θα ήθελα να δω το πνεύμα της τροπολογίας μου παριθμών 77, περί ΦΠΑ. Λέγαμε ότι πολιτισμικά προϊόντα, πολιτιστικά προϊόντα και υπηρεσίες πρέπει να θεωρούνται σαν αγαθά πρώτης ανάγκης. Όταν εξετάζουμε τη διαφοροποιημένη αντιμετώπιση του ΦΠΑ. Ε, αυτό είναι βασικό ζήτημα. Στην Ισπανία η κυβέρνηση αύξησε το ΦΠΑ για πολιτιστικά προϊόντα, θέατρα και κινηματογράφο και ήταν κάτι επιζήμιο για τον τομέα και θα, θέλα, θα ήθελα ή δυνατόν να συμπεριληφθεί αυτή η προοπτική στη συμβιβαστική. Διαφορετικά θα αποσύρω το όνομά μου από τη συμβιβαστική τροπολογία. Α, και όχι μόνο μέσω email να έχουμε επαφή, αλλά θέλουμε και με φυσική παρουσία μια συνάντηση, να συζητήσουμε πρόσωπο με πρόσωπο, όχι μόνο μέσω email αυτά τα σημεία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τρεμόσα και σας ευχαριστώ που είπατε και για την περιφέρειά μου την Ναβάρα. Και όπως το έχουμε ξαναπεί δεν χρειάζεται μόνο να υπάρχουν καλά συστήματα αλλά και καλοί κυβερνώντες για να μπορεί να είναι επιτυχημένη από οικονομική πλευρά μια περιφέρεια. Τώρα εξ των πρασίνων δεν βλέπω κανέναν. Για να δω ποιοι είναι εδώ από το ECR. Κανείς. Από την είναι ο κύριος Κλούτε εδώ. Θέλετε κύριε Κλούτε το λόγο, παρακαλώ. Ναι, ίσως ε, σύντομα. Δεν είμαι με ο σκιώδης από την ομάδα μου και δεν έχω λάβει οδηγίες από τον σκιώδη εισηγητή, αλλά να πω δύο λόγια για θέματα φορολογικής εναρμόνισης. Νομίζω ότι από τα τελευταία χρόνια έχουμε διδαχθεί ότι ο φορολογικός ανταγωνισμό έχει και ε, ένα σαφή αρνητικό αντίκτυπο. Τα έσοδα του κράτους ε, βλέπουμε γιατί ξέρετε στη Γερμανία έχουμε παρόμοια προβλήματα και παρόμοιες δομές ε, μεταξύ των κρατηδίων όπως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο αντίκτυπος λοιπόν είναι ότι πέφτουν οι φορολογικοί συντελεστές και τα έσοδα από τους φόρους και αυτό επίσης συνέβαλε στην χρήση των δημοσιονομικών. Άρα θεωρώ ότι το να περιερίσουμε την αντικτύπω αυτό χρειάζεται μια εναρμόνιση του ελάχιστου φόρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η εναρμόνιση αυτή όταν θέλουμε, αν θέλουμε όπως είπε και ο συνάδελφος, μια εναρμόνιση των φορολογικών συστημάτων, θα πρέπει να κάνουμε κάτι παρόμοιο σε ό,τι αφορά τους ελάχιστους συντελεστές ιδάλλως θα προκληθούν ε, ανισότητες ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό δεν θα συνδράμει στην ενίσχυση της Ένωσης ως μια Ένωση ειρήνης και ισορροπίας και ισότητας στο μυαλό του πολίτη. Δεν μπορώ να σας παρουσιάσω τις λεπτομέρειες του εισηγητή του σκιώδη εισηγητή μας από την ομάδα, γιατί δεν τις γνωρίζω, αλλά νομίζω ότι η βασική ιδέα θα πρέπει να είναι ότι ο φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των... Ε, ο φορολογικός ανταγωνισμός τα τελευταία χρόνια οδήγησε σε, και αυτός στην κρίση, στην βάθμιση της κρίσης. Αυτά ήθελα να σας αναφέρω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Αν δεν θέλει κανένας άλλος ε, το λόγο, το λόγο έχει και πάλι η συγγήτρια. Η κυρία Γκαλπέλης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τους σκιώτες Ε, Σημείωσα πολλά χρήσιμα στοιχεία και φυσικά θα έχουμε συνάντηση την επόμενη εβδομάδα με φυσική παρουσία. Ελπίζω στις 17 Απριλίου να το καταφέρουμε αυτό. Στις 17 Απριλίου θέλω λοιπόν να συγκαλέσω συνάντηση με τους κοιότητες συζήτητες. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχετε και εσείς την εντύπωση ότι η συζήτηση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και που θεωρείτε ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια κοινή θέση. Το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το ξέραμε αυτό, το ξέραμε αυτό εξ αρχής. Η εναρμόνιση, η φορολογική, η φορολογική, τα θέματα φορολογικού ανταγωνισμού, φορολογικής έντρας. Είναι ένα θέμα αυτό το οποίο πολλώνει. Γι' αυτό έχουμε προτείνει αυτό το σύστημα του φορολογικού φιδιού, όπως αποκαλείται. Η κατάσταση είναι παρόμοια με αυτήν πριν από την εισαγωγή του ευρώ. Χρειαζόμαστε έναν ευφυή συντονισμό. Δεν μιλάμε παρά για ένα σύστημα το οποίο θα ελέγχει ποιος είναι ο αντίκτυπος της αύξησης ή της μείωσης των φορολογικών συντελεστών στα διάφορα κράτη, μέλη, τα οποία έχουν διαφορετική δημοσιονομική πολιτική ασφαλώς. Αυτό αποτυπώνεται στην συμβιβαστική τροπολογία που αναφέρεται στο σημείο 15. Εγώ δεν είμαι πολέμιος της φορολογικής εναρμόνισης. Δεν θεωρώ ότι σε μια τέτοια κρίση όμως που απαιτεί τόσο μεγάλη ενέργεια θα πρέπει να δαπανίσουμε πάρα πολύ, μεγάλο, πάρα πολύ χρόνο στην φορολογική εναρμόνιση. Ανεξάρτητα από το θα είναι καλύτερο στο σύστημα ή όχι. Ένα σύστημα όμως το οποίο θα παρακολουθεί τις επιπτώσεις των φορολογικών μέτρων θεωρώ ότι είναι χρήσιμο και θετικό. Αυτό το σύστημα ακριβώς αυτόν τον σκοπό θα εξυπηρετήσει και αυτό αποτυπώνεται σε μια συμβιβαστική πρόταση που έχω καταθέσει. Μετά από μια ισβάτος ανάλυση θα μπορούσαμε να προτείνουμε ένα σύστημα το οποίο ενδεχομένω να, να το αποκαλέσουμε φορολογικό φίδι. Δεν μιλάμε ουσιαστικά για φορολογική εναρμόνιση, αλλά για φορολογική διαφάνεια. Μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο θα καταγράφει την αύξηση και τη μείωση της φορολογίας στα κρατημέλη. Κατανοώ το πρόβλημα το οποίο αναφέρθηκε για τις ανισορροπίες ε, εντός της Ένωσης. η ευρωπαϊκή πολιτική μπορεί να μην προσανατολίζεται 100% στην άρση των ανισορροπιών αυτών, αλλά είμαι βέβαιη ότι με την ε, φορολογική πολιτική βασικό μας καθήκον θα πρέπει να είναι η μείωση έστω των ανισοτήτων αυτών. Ο κύριος Φαμόζα. ανέφερε στο σημείο αυτό ότι υπάρχουν περιφέρειες που έχουν αρμοδιότητα για την επιβολή και την ίσπραξη φόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ασκούνται με πολύ διαφορετικό τρόπο ε, οι εξουσίες διακυβέρνησης διοίκησης είναι πολλές και διαφορετικές οι περιφέρειες. Σε ό,τι αφορά θέματα φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, τα τόνισα τα ζητήματα αυτά. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά. Και θεωρώ ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής είναι σωστή. Στο πλαίσιο αυτό. Έλαβα και γραπτές παρατηρήσεις ε, από τους συναδέλφους. Δεν θα επισέλθω σε αυτές αυτή τη στιγμή. Θα τις συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος, κυρία Γκάλ Και για να ε, ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, να σας πω ότι στις 21 Απριλίου θα γίνει η συζήτηση και η ψηφοφορία και στην ε, Ολομέλεια θα ψηφιστεί το Μάιο το θέμα αυτό. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το σημείο 9 και 10. Το 9 είναι η τροποποίηση του κανονισμού υπαριθμών 653 του 1999 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 93 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής και το θέμα 10 έχει να κάνει με την τροποποίηση του κανονισμού Υπαριθμών 994 του 98 για την ίδρυση σε ορισμένες κατηγορίες ε, οριζόντων κρατικών ενισχύσεων και του κανονισμού υπαριθμών 1370 του 2007 για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και δικές μεταφορές. Θα συζητήσουμε από κοινού τις ε, δύο αυτές εκθέσεις και θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Ντόρφμαν, ο οποίος είναι εισηγητής της δεύτερης έκθεσης. Έχετε το λόγο κύριε Ντόρφμαν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε. Μιλάμε για τον κανονισμό block exemptions. Μία δυνατότητα που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εξαίρεση ε, ορισμένων κατηγοριών από τις ε, υποχρεώσεις αναφοράς. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε ότι θα ήταν σκόπιμη η επέκταση αυτού του κανονισμού για να προβλεφθούν νέες κατηγορίες σε ό,τι αφορά τις εξαιρέσεις αυτές για το πότε δεν είναι απαραίτητη η υποβολή αυτών των εκθέσεων, των αναφορών. Αυτές οι νέες κατηγορίες που προβλέπει και προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο τομέας της πολιτισμικός, ε, πολιτισμικής κληρονομιάς, ε, θέματα μετά από ε, φυσικές καταστροφές. Κατά τρίτον, ο αλληλευτικός τομέας σε ό,τι αφορά τις ενισχύσεις. Οι ενισχύσεις για θέματα καινοτομίας, δασοκομεία και ο τομέας των τροφίμων, παραγωγής τροφίμων, κατά έκτο ε, βιολογικά συστήματα, ερασιτεχνικός αθλητισμός, οι αποκεντρωμένες περιοχές όπως νησιωτικές περιοχές, σε ε, μεταφορές και τα αντιφατικά ε, τα δίκτυα νέας γενιάς. Δεν είμαστε όμως σε διαδικασία συναπόφασης. Κάνουμε μια γνωμοδότηση προς το Συμβούλιο και το Συμβούλιο είναι αυτό το οποίο τελικά θα πρέπει να αποφασίσει για τον νέο κανονισμό αυτό. Στην έκθεσή μου προτείνω κάποιες τροπολογίες και ζητώ αυτές οι κατηγορίες να οριστούν πιο με μεγαλύτερη ακρίβεια. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, θεωρώ ότι καλό θα είναι να συνάδουμε με, τον, ε, με τους στόχους της Ευρώπης 2020 σε ό,τι αφορά τον τεχνικό αθλητισμό. Πολύ καλή εξαίρεση και σκόπιμη σε ό,τι αφορά τις αθλητικές ενώσεις, αλλά όχι σε ό,τι αφορά τα έργα υποδομών στον τομέα των δικτύων ταχείας πρόσβασης, τα ευρυζωνικά δίκτυα, καλό είναι να υπάρχει πρόσβαση στα δικτύα αυτά φυσικά. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε, επειδή παράλληλα γίνονται και εργασίες για ένα κανονισμό για το ευρυπαϊκή Νομοθεσία Προμηθειών, θα πρέπει να κινούμαστε παράλληλα. Και θα πρέπει να υπάρχει φυσικά δίκαιος ανταγωνισμός για την διαδικασία. Ακούγεται, α, φυσικά πρόκειται για ένα δημοκρατικό έλμα το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν συμμετέχει με τη διαδικασία συναπόφασης. Σε ό,τι αφορά τις ενισχύσεις, σε ό,τι αφορά τις ε, ενδεχόμενες άλλες κατηγορίες που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν. Ως κοινοβούλιο προτείνω ότι μιας και δεν συμμετέχουμε στην διαδικασία συναπόφασης, τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια προτείνω να ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώνει σε ό,τι αφορά τον κανονισμό για τις εξαιρέσεις αυτές. Και τέλος υπάρχει ένας άλλος σημαντικός τομέας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαγράψουμε το άρθρο 9 του α, κανονισμού του 2009. που ορίζει τις εξαιρέσεις σε ό,τι αφορά τον τομέα των δημόσιων μεταφορών. Εδώ θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι δημοκρατικής φύσεως. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά τον κανονισμό 1370 του 2007 και το άρθρο 9, έχουμε διαδικασία συναπόφασης. Πώς μπορούμε δηλαδή να αποφασίζουμε με τον κανονισμό αυτό που δεν προβλέπει συναπόφαση για ένα θέμα το οποίο εμπίπτει στα πλαίσια της συναπόφασης. Και οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Μεταφορών είναι αρμόδιοι καθήλυν για τον τομέα αυτό. Άρα θεωρώ ότι θα πρέπει να αντιταχθούμε. Δεν είναι δυνατόν με τον κανονισμό αυτό να τροποποιείται ο 1370 του 2007. Εάν θέλει να αλλάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον 1370, να το κάνει με μια διαδικασία συναπόφασης. και οι συνάδελφοι της Επιτροπής Μεταφορών θα αποφανθούν κατά πόσον πρέπει ή όχι να τροποποιηθεί ή να διαγραφεί το άρθρο 9. Αυτά επί του περιεχομένου, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Thank you very much indeed, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντόρκμαν. Τώρα εξ ονόματος των σοσιαλιστών θα δώσω το λόγο στον κύριο Κούντα, στο σκιώδη συγητή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ και τους δύο συγητές για τη δουλειά τους. Και θα συνεργαστώ με τα χαράς μαζί τους. Για τον κύριο Ντόρμα να πούμε να έχετε δίκιο και θα το πω και για την κυρία Πιετικάινεν που είπε πολύ ξεκάθαρα στην έκθεσή της ότι υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα με το 109 άρθρο να χρησιμοποιηθεί δηλαδή ως νομική βάση και για τους δύο κανονισμούς, αλλά δυστυχώς ε, αυτό είναι και μας δίνει μόνο δικαίωμα διαβούλευσης. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε ε, με το άρθρο 9 που αναφέρεται αν μπορούμε να το ακυρώσουμε. Υπάρχει διαβούλευση τώρα σχετική, αλλά θα τα συζητήσουμε και με τους εισηγητές για να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Καταρχάς τώρα να πω κάποια λόγια για την έκθεση της κυρίας Πιετικάινεν. Πιστεύω ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι πολύ καλή και είναι ένα σημαντικό βήμα για τον εξυγχρονισμό των ε, διαδικασιών των κρατικών ενισχύσεων και για να είναι πιο αποτελεσματική η διαδικασία της συμμόρφωσης από την Κομισιόν. Επίσης βλέπουμε ότι η συνεργασία μεταξύ Κομισιών και Εθνικών ε, Ερευνητικών Συνεδρίων είναι κάτι θετικό και πρέπει να το στηρίξουμε. Ενώ στηρίζω και την ιδέα να έχει τη δυνατότητα η Κομισιόν να λαμβάνει από τους συμμετέχοντες ε, στην αγορά άμεσα όλες τις πληροφορίες, αν οι πληροφορίες που δίνουν τα κρατημέλη δεν επαρκούν βέβαια και νομίζω ότι με αυτό το μέτρο θα αυξηθεί η διαφάνεια. Έκθεση Ντόρφμα τώρα. Και αυτή η έκθεση είναι σημαντική. Όπως είπε, κάποιες κατηγορίες ε, ενισχύσεων για τον πολιτισμό, παραδείγματο χάρη για την αποζημίωση, λόγω φυσικών καταστροφών θα εξαιρούνται. ή βοήθεια σε κάποιες υποδομές κτλ. Και σε ό,τι αφορά την έρευνα ανάπτυξη και ανατομία, συμφωνώ ότι θα πρέπει να εφηγραμμιστούν με τις εμβληματικές πρωτοβουλίες για την Ευρώπη του 2020. Θα πρότεινα πάντως να μην προσπαθήσουμε να είμαστε πάρα πολύ περιοριστικοί, αλλά να ανοίξουμε την πόρτα και για άλλες πρωτοβουλίες για την στρατηγική για την 2020. Τέλος, θα ήθελα να προτείνω και στους δύο εισηγητές να λάβουν υπόψη ε, την ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας. Νομίζω ότι είναι καλύτερο η ψηφοφορία να γίνει πριν τη συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 29 Μαΐου. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα, παρότι πρόκειται για τη δικασία διαβούλευσης, να επηρεάσουμε, έτσι πιστεύω τουλάχιστον, και τις συζητήσεις στο επίπεδο του Συμβουλίου. Προσβλέπω λοιπόν στη συνεργασία μας και σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κούτας και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Καϊνεν την εισηγήτρια του πρώτου φακέλου, της πρώτης ε, έκθεσης. Ευχαριστώ ξεκινήσατε 15 λεπτά νωρίτερα, ίσως και πιο, πιο νωρίς από ό,τι προγραμματιζόταν. Γι' αυτό άργησα. Ήμουνα σε άλλη επιτροπή. Ήμουνα σκιώδης συγγήτρια για άλλη έκθεση. Εν πάση περιπτώσει. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση εδώ και είναι καλό. Όπως γνωρίζουμε όλοι, ο κανονισμός με τον οποίο ασχολούμαστε βάσει το άρθρο 107 και 108 των συνθήκων που καθορίζουν τους ε, κανόνες για τα κράτη-μέλη και τους ορισμούς της κρατικής ενίσχυσης και τους λόγους χορηγήσεως της ενίσχυσης και πώς μπορεί να μην δημιουργεί στρέβλωση ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά αυτή η ενίσχυση και τις διάφορες διαδικαστικές αρχές που διέπουν την όλη διαδικασία και πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζεται ότι τα κράτη-μέλη συμμορφώνονται με τον κανονισμό. Αυτό είναι το θέμα μας λοιπόν. Ο κανονισμός αυτός δεν τροποποιήθηκε σημαντικά από όταν εγκρίθηκε αρχικά. Οι αλλαγές ίσως φαίνονται τεχνικής φύσεως Εξαρτάται όμως η εφαρμογή μιας αρχής για να κάνει τη διαφορά. Και ήρθε η ώρα των αλλαγών. Το ανέφερε και στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή περί εξυγχρονισμού της κρατικής ενίσχυσης. Στόχος του τους είναι η δημόσια χρηματοδότηση να προσαρμοστεί με τους στόχους του 2020. Να χρησιμοποιηθεί λοιπόν κατάλληλη κρατική ενίσχυση για καινοτόμο ανάπτυξη με κοινωνική συμπερίληψη των πάντων. Έχουμε δημοσιονομικούς περιορισμούς όμως ταυτόχρονα. Και θέλουμε εξυγίανση του προπολογισμού. Να χρησιμοποιούμε σωστά τα χρήματα με άλλα λόγια. Άρα πρέπει να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων. Ποιο ήταν το πρόβλημα μέχρι τώρα. Οι διαδικασίες και ερμηνείες πίκυλαν, πικίλαν μάλλον στις διάφορες χώρες. Δεν δόθηκε κατάλληλη σημασία στα μέτρα που έδιναν τα σωστά αποτελέσματα και δεν υπήρχαν τα κατάλληλα εργαλεία για να εντοπίσουμε τους μεγάλους στόχους και τα μεγάλα προβλήματα και πού δημιουργούνται στρεβλώσεις από την κρατική ενίσχυση. Ας πούμε ναυπηγεία παραδείγματος χάρη. Ο ανταγωνισμό εκεί ήταν πολύ στρεβλό όσον αφορά την αφήγηση σκαφών και τι επισκευέ του, λόγω κρατικών ενισχύσεων. δι, διτό στόχο έχουν οι βελτιώσεις για να βελτιώσουμε την επεξεργασία των καταγγελιών. Μέχρι τώρα δεν είχαμε σωστό έλεγχο. Τι γινόταν. Μπορούσε, καθ... μάλλον μπορεί τώρα ο καθένας να καταγγείλει κρατική ενίσχυση και προβλήματα, ε, να απευθυνθεί προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακόμα και αβάσιμες καταγγελίες μπορούσαν να υποβληθούν. Ας πούμε θα μπορούσαν και κάποιοι ανταγωνιστές οι οποίοι δεν ήταν ευχαριστημένοι και ήταν σε δύσκολη θέση να κάνουν καταγγελίες για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό. Και μέχρι τώρα δεν γινόταν σωστές προσπάθειες τα χρήματα να πηγαίνουν για το σωστό σκοπό. Θέλουμε λοιπόν να βελτιώσουμε την επεξεργασία των καταγγελιών και των διαμαρτυριών. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει περισσότερους πόρους για να ερευνά τη σοβαρότητα των ε, υποθέσεων. Να βλέπει ποιε είναι σοβαρές και ποιες όχι. Και όταν υποβάλλεται μια καταγγελία στο μέλλον θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά κάποιο ελάχιστο αριθμό πληροφοριών πρέπει κανείς να μπορεί να αποδείξει ότι έχει βάσιμους λόγους για την καταγγελία και ότι είσαι εμπλεκόμενο μέρος και επηρεάζεσαι. Και πρέπει να αναφέρεις ποιες είναι οι καζόμενες καταχρήσεις της κρατικής ενίσχυσης. Θέλουμε ταχεία αντιμετώπιση, fast track των καταγγελιών. Δηλαδή, δεν πρέπει να πάρει επίσημα απόφαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν δεν έχουν δοθεί σωστές πληροφορίες. Και όταν είναι σαφές ότι δεν υπάρχει παράβαση των κανόνων των κρατικών περιενισχύσεων. περί ενισχύσεων. Έτσι επιταχύνεται η διαδικασία. Δεν ξεκινά καν η διαδικασία διότι ε, εκ των πραγμάτων διαπιστώνεται ότι δεν είναι βάσιμη η καταγγελία. Άλλη προσπάθεια. Πώς εφαρμόζονται οι κανόνες σε εθνικό επίπεδο, να ξέρουμε ακριβώς πώς εφαρμόζονται. Πρόταση. να έχει πιο καλά και πιο πρακτικά εργαλεία για να υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, τα εθνικά δικαστήρια τις αποφάσεις που λαμβάνουν. Μπορεί να παρέχει πληροφορίες απευθείας στα δικαστήρια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σχετικά με το σκοπό χορηγήσεως κρατικών ενισχύσεων, τον αποδεκτό, μπορεί να προσφέρει στα εθνικά δικαστήρια η Κομισιόν. Πολύ ευπρόσδεκτη προσέγγιση αυτή. Θέλουμε αποτελεσματική συλλογή πληροφοριών. Νέο σημαντικό στοιχείο προτείνεται σχετικά με αυτό. Πληροφορίες, εργαλεία για τη συλλογή πληροφοριών που αφορούν την αγορά θα μπορεί να απαιτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφορίες από φορείς πέραν των κρατών μελών, εκτός των κρατών μελών. Άρα πιο γρήγορα και αποτελεσματικά θα συλλέγονται οι πληροφορίες σχετικά με τις μεγάλες υποθέσεις, τις σημαντικές υποθέσεις. Όταν τα κράτη-μέλη ίσως διστάζουν να δώσουν πληροφορίες γρήγορα, ίσως να μην θέλουν να δώσουν πληροφορίες καθόλου. Έτσι η έρευνα θα διενεργείται ακριβέστερα, ταχύτερα, με καλύτερη μέθοδο. Είναι καλή και η εισαγωγή κυρώσεων, την υποστηρίζω. Όταν χορηγούνται λανθασμένες πληροφορίες και όταν δεν ακολουθούνται οι σωστές διαδικασίες, να επιβάλλονται ποινές. τίθενται ένα-δύο άλλα θέματα που σχετίζονται κάπως με τις κρατικές ενισχύσεις και τα συναφή ζητήματα. Δηλαδή, πώς ερμηνεύουν τους κανόνες τα κράτη-μέλη. Δεν γίνονται δοκιμέ όσον αφορά την αγορά και πώ επηρεάζεται από τι διάφορε ερμηνείε. Το τυπτογενή τομέα αφορά περισσότερο αυτό. στο ε, κατά πόσο υπάρχει μια αγορά, αν ισχύουν οι κανόνες περικρατικών μια αγορά, ας πούμε ΜΚΟ, που προσφέρουν υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία, μεγάλα ιδρύματα που στον τομέα της υγείας. Είναι διοικητικό άχθος να εξετάζονται αυτές οι περιπτώσεις στα κράτη-μέλη και απ' την άλλη ίσως να ενθαρρύνει υποβολή καταγγελιών που δεν χρειάζονται. Και σε περίπτωση κοινωνικών προβλημάτων ίσως να εμποδίζουμε τη χρήση δημοσίων πόρων για τον τιτογενή τομέα που προσπαθεί να υποστηρίξει τους πολίτες. Προτείνω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιμείνει τα κράτη-μέλη να διευκρινίσουν ποια είναι η κατάσταση να γίνει μια αξιολόγηση των αγορών, να γίνει δοκιμή αγορών. Πού εφαρμόζονται οι κανόνες για κρατική ενίσχυση στα κρατη τα μεγάλα θέματα πρέπει να είμαστε πολύ πιο αυστηροί. Για άλλε περιπτώσεις, όταν μιλάμε για τον τριτογενή τομέα, την κοινωνία των πολιτών, να κάνουμε διαχωρισμό να εφαρμόσουν πιο χαλαρά οι κανόνες περικρατικής ε, ενίσχυσης. Αυτό το δρόμο διάλεξα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και προσβλέπω στα σχόλιά σας και τις προτάσεις σας για περαιτέρω εξέλιξη των εργασιών. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πίτη ευχαριστώ κύριε Κούτας που είναι εισηγητής και για τις δύο εκθέσεις. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάτι στα σχόλια της κυρίας Πιτικάνεν. Ευχαριστώ. Εκ μέρου τη Άλτε, η κυρία Ινβέλτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Η Σάρων Μπόλη μου ζήτησε, η οποία είναι σκιώδη γήτρια από τι εκθέσει Κάινεν, μου ζήτησε να αναγνώσω ένα κείμενο που έχει ετοιμάσει. Αλλά πρώτα θα κάνω και προσωπικέ παρατηρήσει για την έκθεση Dorfman, τη οποία είμαι εγώ σκιώδη εισηγήτρια. Θέλω να σα ευχαριστήσω λοιπόν πρώτα απ' όλα για την έκθεση, η οποία είναι πάρα πολύ περιεκτική, ξεκάθαρη. Και πρέπει να πω ότι και το έχω ξαναπεί, σε γενικέ γραμμέ ε, δεν είμαι τόσο σίγουροι για το κατά πόσο πρέπει να ανοίγουμε συνεχώς το πεδίο εφαρμογή με κανονισμούς ε, ε, περί εξαιρέσεων. Ο στόχος φαίνεται καλός, αλλά πρέπει να προσέξουμε πολύ καλύτερα την πρακτική εφαρμογή αυτών των εξαιρέσεων, γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι κρατικών ενισχύσεων που δεν αιτιολογείται, είτε δεν αιτιολογείται επαρκώ, είτε καθόλου. Και όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μα πρώτου σκεφτούμε να ε, διευρύνουμε το πεδίο των εξαιρέσεων ε, στους κανονισμούς. ό,τι αφορά τώρα το να προσπαθήσουμε να ψαρέψουμε το μεγάλο ψάρι, ε, συμφωνώ ε, με το στόχο επί της αρχής, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει και τα μικρά ψάρια να τα αφήσουμε ε, γιατί και αυτά μπορούν να επηρεάσουν την αγορά. Να μην τα παραγνωρίσουμε δηλαδή εντελώς από την αρχή και από την έννοια αυτή καλωσορίζω και τις προτάσεις του κυρίου Ντόρφμαν για παράδειγμα σε ό,τι αφορά το καθορισμό ξεκάθαρων κριτηρίων για τις εξαιρέσεις. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ καλό για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. και οι τροπολογίες 8 και 9 του κ. Ντόρφμαν για του κανόνες περί δημοσίων προμηθειών για να υπάρχει ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού είναι πολύ σημαντικές και τι ε, ε, επικροτώ. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας το γεγονό ότι οι κρατικές ενισχύσει πρέπει να παραμένουν πάντοτε εξαίρεση, να είναι κάτι προσωρινό πάντα. Και δεν θα πρέπει έτσι κάπως με λαθάνοντα τρόπο ή φέρποντα τρόπο να γίνει μόνιμη κατάσταση. Επίσης δεν έχω ξετρελαθεί, ακόμη τουλάχιστον, ε, θα το δω βέβαια, το θέμα της τροπολίας 6, 6 όπου προτείνεται ε, να μην υπάρχει νοποίηση των ε, κρατικών ισχυρών, υπάρχει συγχρηματοδότηση, γιατί λέτε ότι ήδη υπάρχει έλεγχος, αλλά δεν είμαι πεπισμένη γι' αυτό. Ο έλεγχος δεν νομίζω ότι είναι 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεσματικός και γι' αυτό πριν κάνουμε παραπάνω προτάσεις να τα δούμε όλα αυτά. Τέλος, συμφωνώ και μαζί σας αλλά και με την κυρία Πιετικά είναι το δημοκρατικό έλλειμμα και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι σίγουρα εύκολα θα υπάρξει συνένεση γι' αυτό στην Επιτροπή μας. Τώρα, η συνάδελφός μας, η Σάρουν που δυστυχώς είναι στο Δουβλίνο σήμερα για να μιλήσει στο άτυπο συμβούλιο του ΕΚΟΦΗΝ μεταξύ άλλων, ε, μου έδωσε να διαβάσω ένα κείμενο, αν με επιτρέπετε τώρα. Λέει λοιπόν ότι ο στόχος αυτού του κανονισμού για την έκθεση ποιητικά είναι συγκεκριμένα αναφέρεται, είναι να βελτιωθεί ο κανονισμός ε, του 99 για να είναι μικρότερο ο χρόνο τη διερεύνηση ε, καταγγελιών για κρατικέ ενισχύσει, για να είναι δηλαδή γνήσιε οι καταγγελίε, ε, να επιβεβαιωθεί και να αυξηθεί η διαφάνεια τη όλη διαδικασία, όπω και η συγγήτρια. Συμφωνώ με αυτό το οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μεγαλύτερο μέρο, γιατί είναι ε, λογικέ απαιτούμενε τροποποίησει του εφιστάμενου κανονισμού. Βέβαια, θα πρέπει να επιμείνουμε ότι οι καταγγελίε θα πρέπει να είναι βασισμένε σε στοιχεία, σε αποδείξει, να και σε ό,τι αφορά δηλαδή την ενημέρωση για το ενδιαφερόμενο μέρο ε, και την ε, καταγγελία θα πρέπει οι πληροφορίε να γνωστοποιούνται. Σε ό,τι αφορά τώρα το market testing στην τροπολογία, δεν είναι ενδιαφέρον ω ιδέα και θα ήθελα να ακούσω περισσότερε λεπτομέρειε. Η αναφορά τώρα στο πραγματικό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά και το πώς αυτό ε, αντιστοιχίζεται με την εντολή της Κομισιόν. Είναι κάτι που με ανησύχησε λίγο και ίσως θα πρέπει να το δούμε στην ε, με τους Σκιώδη. Στην αρχή ε, η, της εκπαικοδομητικής ε, συμμετοχής των Σκιώδων και όχι μόνο ατομικά στην τροπολογία 8 είναι καλή ιδέα και ίσως θα πρέπει η Κομισιόν να ε, παράγει και να υποβάλει στο Κοινοβούλιο ενδιάμεσες εκθέσεις. Για τη διαφάνεια όχι μόνο η Κομισιό θα πρέπει να δημοσιεύει τα αποτελέσματα των καταγγελιών για κρατικέ ενισχύσει στην επίσημη εφημερίδα, όπω γίνεται με τον ισχύοντα κανονισμό, αλλά θα πρέπει να τι δημοσιεύει και στην gmail.com, ε, στην ιστοσελίδα τη DigiCom. Βρύτερα ε, τώρα, σε ό,τι αφορά το ρόλο του Κοινοβουλίου, στην Επιτροπή μας δίνω μάχες και με την Επιτροπή Τραν, γιατί στο άρθρο 2 διαγράφεται ένα άρθρο από τον ε, κώδικα περί συναπόφασης. Είναι μια ανησυχητική τάση με, το, με τη μάχη αυτή που γίνεται για τις αρμοδιότητες. Μπορεί να θεωρεί θεμητή την κίνηση αυτή το, η Κομισιόν, αλλά εμεί θα πρέπει να πιέσουμε να υπάρχει μεγαλύτερο έλεγχος και όχι να χάσουμε ένα κομμάτι Τροπολογία 3 και τροπολογία 10 Ντόρφμαν. Σημαντικές. Ζητώ συγγνώμη που δεν μπορώ να είμαι εδώ σήμερα. Αλλά θα τα πούμε στην συνεδρία των σκιωδών. Σα ευχαριστώ πολύ, κυρία Ίντφελτ. Τώρα, εξ ονομάτων των Πρασίνων, το λόγο έχει ο κύριος Μπέσετ που είναι αρμόδιος για τις δύο εκθέσεις. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να κάνω κάποια σχόλια γρήγορα. Εν γέννη, πιστεύουμε, όπως και η συγγήτρια άλλωστε, η κυρία Πίτη ότι ο προτινόμενος κανονισμός ακολουθεί σωστή κατεύθυνση. Θα επιτρέψει βελτίωση και εξορθολογισμό των διαθεσίμων εργαλείων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μειώνοντας το διοικητικό άχθος των κρατών μελών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις. Είμαστε υπέρ των προβλεπωμένων εργαλείων ενημέρωσης και πληροφόρησης για την αγορά και των ερευνών κατά οικονομικούς τομείς. Ελπίζουμε να εφαρμοστεί με δυναμικό τρόπο αυτό. Κυρίως για τον τραπεζικό τομέα που έχει λάβει άνευ προηγουμένου κρατικές ενισχύσεις από την αρχή της κρίσεως. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια για το σχέδιο έκθεσης. Το υποστηρίζουμε ανεπιφύλακτα κυρίως τις τροπολογίες 8, 14, 15 που επεκτείνουν τι ε, τις έρευνες, τις ε, που μπορεί να διενεργούνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το για την έκθεση Dorfman που την έκθεση το οποίο υποστηρίζουμε ανεπιφύλακτα. Είμαστε υπέρ τη συμπεριλήψεως των προβλεπωμένων πρωτοβουλειών στα πλαίσια της στρατηγικής 2020 σαν πλαίσιο αναφοράς για την αξιολόγηση του βασίμου των κρατικών ενισχύσεων και της υποστήριξης της καινοτομίας. Είμαστε εξίσου υπέρ της επιλογής του εισηγητού όσον αφορά την αντιμετώπιση των κοινοποίησεων στις χερσαίες μεταφορές. Εξάλλου, Είμαστε υπέρ, πολύ υπέρ της τροπολογίας 10 που θέλει να καλύψει το δημοκρατικό έλλειμμα της νομικής βάσης του κανονισμού, δηλαδή το άρθρο 109 της συνθήκης. Συνεπώς καλούμε το Κοινοβούλιο να χρησιμοποιήσει τη ρήτρα πασαρέλας που προβλέπεται στο άρθρο 48.7 της συνθήκης που επιτρέπει με ομοφωνία το Συμβούλιο μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κατόπιν αιτήματος θεσμικού οργάνου να περάσει την έγκριση του νομικού κειμένου με ειδική διαδικασία χωρίς να περάσει από κανονική αναθεώρηση της ε, συνθήκης. Θέλουμε και στις δύο εκθέσεις Dorfman και Επίτη Κάνεν να εκφράσει σαφής βούλησης να πάμε προς χρήση ρήτρας πασαρέλας και να ζητήσουμε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να το υλοποιήσει. Αυτό ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπέσετ, εξ ονόματος της ΓΚΟΕ, να ακούσουμε τον κύριο Κλούτα, που είναι εισηγητής και για τις δύο εκθέσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με αυτά που ακούσαμε έως τώρα. Μία παρατηρήση επί της αρχής όμως να κάνω. Δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε η συνάδελφος Ιντσφέλτ. Επί της αρχής σήμερα δεν εγκρίνονται οι κρατικές ενισχύσεις και όπου εγκρίνονται υπάρχουν εξαιρέσεις. Εγώ προσωπικά θα προτιμούσα να υπάρχει ένα σαφή διαχωρισμό. Υπάρχουν τομεί στου οποίου προβλέπονται κρατικέ ενισχύσει, όχι εξαιρέσει, ορίζονται με σαφήνεια. Αυτό θεωρώ ότι είναι ιδεολογικό ζήτημα το οποίο δεν πρόκειται να το λύσουμε σήμερα για τις συγκεκριμένε προτάσεις και για τις δύο εκθέσεις. Τις υποστηρίζουμε και πρόκειται να τις υποστηρίξουμε. Μία παρατηρήση για την έκθεση Dorfman. Ο κύριος Dorfman είχε προτείνει κάποιες πρόσθετες εξαιρέσεις. Δεν είναι σαφές για μένα στη Γερμανία σε ό,τι αφορά την νηπιακή και την προνηπιακή και τη σχολική εκπαίδευση έχουμε μια τάση ιδιωτικοποίηση και αυτό επηρεάζει τις ενισχύσεις και αυτό θεωρώ ότι ενδεχομένως να επηρεάζει το κατά πόσον θα πρέπει να θεωρηθούν τομείς εξαίρεσης ή όχι αυτοί οι τομείς, αλλά αυτό ίσως να είναι κάτι κατεξοχή γερμανικό για την έκθεση τι ναι. Υποστηρίζουμε αυτά που ακούσαμε για το θέμα της διαφάνειας και θεωρώ ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγχει τις μεμονωμένες επιχειρήσεις. Αν δεν υπάρχουν ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες. Αλλά αυτό έχει και συνέπειες σε ό,τι αφορά την ε, αρμοδιότητα και την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό θα πρέπει να επηρεάσει και την ισορροπία από την πλευρά του ελέγχου. Θα πρέπει να σκεφτούμε με ποιον τρόπο ελέγχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα πρέπει ίσω να εκχωρήσει αρμοδιότητε ελέγχου στο Κοινοβούλιο για να μην υπάρχει κατάχρηση εξουσία ενδεχομένω από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να μην υπάρχει καν αυτή η δυνατότητα. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια σαφή ρύθμιση σε ό,τι αφορά τον έλεγχο τώρα, σε ό,τι αφορά τον ρόλο του Κοινοβουλίου. Εν γέννη, υποστηρίζω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι και θα ήθελα να υποστηρίξω επίσης αυτά που είπε η κυρία ποιοτικά είναι για το θέμα της κοινωνίας των πολιτών. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά σκόπιμο ο τομέας αυτός που ως τώρα δεν έχει παίξει μεγάλο ρόλο στην ομοθεσία της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης να λάβει μεγαλύτερη σημασία, να λάβει μια οποιοδήποτε σημασία στην ομοθεσία μέσω της διαδικασίας αυτή. Αυτές οι παρτρήσεις μου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κλούτε, λέει ο Πρόεδρος και τώρα θα δώσω το λόγο στους συζητητές. Καταρχάς, στην κυρία Πιετικάινεν, αν θέλει να σχολιάσει αυτά που πάνε συνάδελφοι. I think, uh, thank all of you for uh, your very... Σας ευχαριστώ όλους για τα καλά επικοδομητικά σας σχόλια. Σημειώνω όντως όσα υπόθηκαν. και ε, κάποια άλλα θέματα θα συζητήσουμε με τους σκιώδεις και να δούμε από πού θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ κύριε Πίτη Κάιναν. Να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Ντόρφμαν τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους και συζητητές για την επικοδομητική συνεργασία και την πρόσβαση και την ε, ε, προσέγγιση στην έκθεση. Νομίζω ότι μετά από αυτά που ακούσαμε δεν πρόκειται να υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψεων σε ό,τι αφορά αυτά που είπε ο κύριος Κλούτε τώρα για το ποιε εξαιρέσεις ε, ενδεχομένως να έχουν νόημα, μπορούμε φυσικά να τα συζητήσουμε αυτά. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Κούτας και αυτά που είπε για το χρονοδιάγραμμα, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε. αν είναι καλύτερο για τη θέση του Κοινοβουλίου να υπάρξει μια αναβολή. Ή αντιθέτως αν θέλουμε... Μάλλον αν θέλουμε να επηρεάσουμε το Συμβούλιο θεωρώ ότι όλα αυτά είναι εφικτά και ότι είναι και κάτι το θεμητό αυτό το οποίο θα πρέπει να επιδιώξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντόφμα, λέει ο Πρόεδρος. Να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογίων είναι η 30 Απριλίου. 27 και 28 Μαΐου θα εξετάσουμε τις τροπολογίες. Στην Επιτροπή μας θα ψηφίσουμε στις 6 Ιουνίου και στην Ολομέλεια θα ψηφιστεί η έκθεση τον Ιούλιο. Δεν υπάρχουν άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Να σας ανακοινώσω ότι η προσοχή συνεδρίαση θα λάβει χώρα την Τετάρτη 24 Απριλίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι και από τις 3 το απόγευμα μέχρι τις 6.30. Καθώς και την 5η 25 Απριλίου από τις 9 μέχρι τις 12.30 το πρωί. Σας ευχαριστώ πολύ και τα λέμε λοιπόν σύντομα.